Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας βάσει της ημερησίας διάταξης, η οποία προβλέπει το σημείο 10, απαλλαγή 2010 για τους οργανισμούς. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Μονίκα Λουίζα Μάκοβεϊ που θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Η Στάλφος Μακοβέη έχει το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για το ότι αναλάβατε πρόεδρος μας. Θα είμαι συντομότατη, διότι έχουμε μια ώρα να ακούσουμε τους διάφορους οργανισμούς και μετά να θέσουμε ερωτήσεις. Καλωσορίζω αυτή την ανταλλαγή απόψεων που διεξάγεται με το ελεκτικό συνέδριο. Έχουμε κύριο Γκαλέα από το ελεκτικό συνέδριο στο τμήμα με τα Έχουμε τον κύριο Πάτρικ Γκουντού, τον διευθυντή της, Ευ... της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας Αερομεταφορών και την κυρία Μανουέλα Τόμασιν που είναι ε, ε, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Θαλασσίων Μεταφορών. Να δώσω κάποιες πληροφορίες στους συναδέλφους. Δίνουμε απαλλαγέ σε 24 αποκεντρωμένου οργανισμού, άλλου δύο παραπάνω από πέρσι, δύο παραπάνω φέτο είναι η Europol και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Εργάζομαι, επεξεργάζομαι μαζί με τη γραμματεία τη εκθέση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμε μέσα Φεβρουαρίου. Η πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή σχεδιάζεται για τις 29 Φεβρουαρίου και η υποθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 5 Μαρτίου. Εν γέννη ε, έχουμε παρατήσει κάποια προβλήματα στον τομέα των προμηθειών, των μεταφορών. Θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι εκπληκτικό αλλά δεν αναφέρει κανένα πρόβλημα το ελεκτικό συνέδριο σαν αφορά τις μεταφορές. Ε, βρήκαμε προβλήματα και με τους ανθρωπίνους πόρους, την ανεξαρτησία του υπευθύνου για τα λογιστικά αυτή είναι οι τομεί που σχετίζονται με όλες τις υπηρεσίες, του οργανισμούς. Και ευχαριστώ και θα πρέπει να δώσω ευχαριστώ που δόθηκε συνέχεια στο ερωτηματολόγιο του στο λεκτικό συνέδριο για τις υπηρεσίες, του οργανισμούς. Ε, λάβαμε απαντήσεις, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι πολύ ενημερωτικέ και βασικά δεν συλλέγουν πολλές πληροφορίε μετά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που λάβαμε, δεν λάβαμε συγκεκριμένες ε, αντίστοιχες απαντήσεις. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε ε, μια λύση για τη συλλογή πληροφοριών, να τις λάβουμε από το ελεκτικό συνέδριο. Δράτω με της ευκαιρίας να ζητήσω να μας δώσει το ελεκτικό συνέδριο αυτή την έκθεση για τη βαθμολόγηση Benchmark Report. Είναι στη 17η εκδοχή το κείμενο. Τώρα δεν ξέρω τι είναι η 19η, 20η. Ζητήσαμε εμεί το σχέδιο κειμένου ως είχε όταν το ζητήσαμε. Το ζητάμε και τώρα, όσοι έχει τώρα. Σταματώ εδώ και καλό θα ήταν να ακούσουμε από τους ανεξάρτητες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κυρία Μακοβάη. Έχουμε τον εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκό Ορισμό Ασφάλεια Αεροπορία και τον Ευρωπαϊκό Ορισμό για να Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ο κύριος Πάτρικ Κουντού είναι ο πρώτος, τον οποίο θα δώσω το λόγο. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Συγήτρια, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Μεταφορών, που είναι σημαντικός φορέας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη και νομίζω ότι όλοι ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Για να παρουσιάσω εν συντομία τον οργανισμό μας, θα ήθελα να σας πω ότι αυτός ο οργανισμός έχει έδρα την κολονία, έχει πάνω από 600 εργαζομένους, Μεγάλο ποσοστό είναι εμπειρογνώμονες για τις αερομεταφορές, πολλοί πιλότοι ε, και πιλότοι δοκιμών, πολλοί μηχανικοί, ειδικοί σε όλες τους τομείς που αφορούν την αεροναυτιλία και όπως γνωρίζετε, εφόσον μας δώσατε αυτή την αποστολή, είμαστε υπεύθυνοι τώρα για την ε, ασφάλεια όλων των τομέων των αερομεταφορών, από αεροσκάφη μέχρι αεροδρόμια. Αυτός ο οργανισμός χαρακτηρίζεται από επιχειρησιακά καθήκοντα που αντιμετωπίζονται καθημερινά για να αγγιθούμε την ασφάλεια των αερομεταφορών. Να σας δώσω ένα μοναδικό παράδειγμα πρόσφατο. Σίγουρα θα ακούσατε να γίνεται λόγος για τι, τι κάναμε την Παρασκευή. Αναθέσαμε Ε, μια προσπάθεια γιατί πρέπει να διορθωθούν κάποια προβλήματα που έχει το Airbus A380 στη σταυτερά του. Ε, υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζονται καθημερινά σε όλους τους στόλους των αεροσκαφών. Κάνουμε ελέγχους. Είμαστε μοναδικοί υπεύθυνοι στην Ευρώπη για την πιστοποίηση των αεροσκαφών. Αναλάβαμε αυτό το καθήκον ε, έναντι όλων των κρατών μελών συντάσσουμε όλους τους κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια των αερομεταφορών και προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους διάφορους κανόνες προς έγκριση. Ε, εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίζουμε την ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων στα διάφορα κράτη-μέλη. Και τέλος, και δεν είναι ασήμαντο, εδώ και δύο χρόνια ε, καθορίζουμε και παρακολουθούμε το σχέδιο ασφαλείας αερομεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα σχέδιο δράσης αυτό, υψηλού επίπεδου, που έχει σαν στόχο τη μείωση των βασικών κινδύνων των αερομεταφορών ε, που αφορούν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Των κοινών προβλημάτων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κλείσω τη σύντομη παρουσίαση, συνεχώς προσπαθούμε να προοδεύουμε ε, και Έχουμε το ISO 9001 του 2008, πιστοποίηση ISO, όσον αφορά τις δραστηριότητε της υπηρεσίας μας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας Αερομεταφορών και είμαστε ο μόνος οργανισμός που έχει αυτή την πιστοποίηση ISO 9001 για όλες τις δραστηριότητε μας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το τμήμα εσωτερικού ελέγχου μας εξίσου έχει πιστοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο από την ΙΦΑΣΗ. Ε, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Διευθυντά κύριε Μποκού. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μανουέλα Τομασίνη από την ΕΜΖΑ, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Παρακαλώ. Ε, thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγγήτρια, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, αγαπητοί συνάδελφοι από τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα απ' όλα σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ο Ασκόν ε, Χρέη Γενικό Διευθυντή δεν μπόρεσε να έρθει στη σημαντική αυτή συνάντηση γιατί είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα γνωρίζετε τι έχει συμβεί στην Ιταλία με το Κώστα Κονκόρντια. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί την πλήρη προσοχή και πλήρη ενασχόληση του Γενικού μας Διευθυντή. Να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση. Πάντοτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπιστευόταν ε, την ΕΜΣΑ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και βέβαια είμαι διατεθειμένη να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που τυχόν έχετε για την διαχείριση του 2010. Γνωρίζετε ότι η ΕΜΣΑ δημιουργήθηκε το 2002 μετά το ατύχημα με, την, με το πλοίο Έρικα. Και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε ήταν για την βελτίωση τη ασφάλεια ε, στη θάλασσα, βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντο επίση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καθήκοντα τη υπηρεσία ε, σε, δύο, ε, σε τέσσερις βασικούς τομείς υποδιαιρούνται, σύμφωνα και με την νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα βοηθούμε την Κομισιόν να παρακολουθεί την υλοποίηση της ε, κοινοτικής νομοθεσίας ε, στους τομείς της ασφάλειας της θάλασσας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Δεύτερον, αναπτύσσουμε και ε, ασκούμε τις διάφορες θαλάσσιες δυνατότητες, SafeNet για την ανείχνευση σκαφών και εμπειρευμάτων, φορτίων, ένα άλλο κέντρο δεδομένων ώστε ε, να μπορούμε να ανοιχνεύουμε τα πλοία ευκαιρία και το τέτη με σημαία ε, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το τέτη. Επίσης έχουμε ένα σύστημα για την ετοιμότητα και τη δυνατότητα αντίδρασης και κινητοποίηση στη θάλασσα και μια άλλη υπηρεσία, το CleanSynet, για με στόχο να προστατεύσουμε αποτελεσματικά και από τη ρήπανση λόγω σκαφών τις ακτές μας. Επίσης παρέχουμε τεχνικές επιστημονικές συμβουλές ε, στην Κομισιόν στους σχετικούς τομείς αρμοδιότητάς μας. Σε τον χρόνο νέα καθήκοντα αναλάβαμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ό,τι αφορά ε, την τροποποίηση και του καταστατικού του οργανισμού μας. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν σε ένα δυναμικό περιβάλλον, να εκτελέσουμε σε πολύ στενά και προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα τις, ε, αποστολή αποστολές που μας αναθέτουν τα κρατημέλη και η Κομισιονά. στο 2010 που είναι και ο βασικό στόχο αυτή τη ακρόαση. Ίσως έχετε παρατηρήσει ή διαβάσει στα έγγραφα για την ΕΜΣΑ, Όπω συνήθω ο στόχο μα είναι η καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που μα εκχωρεί η Δημοσιονομική Αρχή. Σε ό,τι αφορά το καταστατικό μα προσωπικό, κλείσαμε τη χρονιά με πολύ μικρά ποσοστά κενών θέσεων, 2% μόνο, 96 θέσεις ε, ε, ε στις 100 ε, είναι κατηλημένες. Η υπηρεσία μας πέτυχε το στόχο του 98% επίσης της εκτέλεσης ε, των πιστώσεων πληρωμών και 98% των πιστώσεων αλήψεων υποχρεώσεων και ένα συν 4% για τις υποχρεώσεις και συν 8% με τις, ε, για τις πληρωμές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα μέτρα επίση για την καταπολέμηση της ρήπανσης τα παρουσιάσαμε, παρουσιάσαμε τα πολύ θετικά μας αποτελέσματα. Τώρα μεταφορές και δεσμεύσεις αποστεριώρη, ε, χάρη στον πολύ αποτελεσματικό εσωτερικό μηχανισμό που έχουμε μετά και από τις πολύ χρήσιμες συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και των ελεκτικού συνέδριου τα προηγούμενα χρόνια, ελέγξαμε την κατάσταση. Το 2015 ε, μόνο ήταν οι υποχρεώσεις ε, στεριόρι, πολύ μεγάλο επίτευγμα. Κάναμε 38 μεταφορές, αλλά πρέπει να σας πω ότι το 2011 μόνο 16 καταφέραμε να κάνουμε. Άρα πολύ θετική η τάση για την υπηρεσία μας. Πολύ μας ενδιαφέρουν οι συστάσεις και υποδείξεις ε, των αρχών της απαλλαγής και φυσικά και του ελεγκτικού συνεδρίου. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς ε, τις επιδόσεις μας ό,τι αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα. Εν συντομία, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε εκπληρώσει ένα πολύ σημαντικό στόχο το 2010. Εγκρίναμε δηλαδή την πενταετή μας στρατηγική μετά από τις υποδείξεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. για πολιετή προγραμματισμό έχουμε κάποιους βασικούς δείκτες επιδόσεων για να μετρήσουμε τις δραστηριότητές μας. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και στο πρόγραμμα εργασίας μας και στα ημετήσια μας έκθεση. Αναθεωρήσαμε επίσης τις εσωτερικές μας διαδικασίες εξασφαλίζοντας ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα σε, όλη την, όλο το φάσμα της οικονομικής μας διαδικασίας. Επίσης, καταφέραμε να υλοποιήσουμε μια σειρά συστάσεων σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του accounting officer Έχουμε ξαναδεί και αν είναι αρκετά διαφανής η, εθνική μας, η ετήσια μας έκθεση. Βλέπουμε και τα διάφορα εθνικά παραρτήματα, διαδικασίες διαπραγματεύσεων και τα οι αποστεριώρες δεσμεύσεις. Όλα αυτά έχουμε περιλάβει πλέον στην ετήσια μας έκθεση. Επίσης το ετήσιο πρόγραμμα το αναθεωρήσαμε για να είναι πιο διαφανές και να αποτελεί τη βάση των αποφάσεων που θα λαμβάνουμε σε όλες τις δικασίες προμηθειών. Επικεντρωθήκαμε όπως πάντα στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και ολοκληρώνοντας να σας πω κάποια αριθμητικά στοιχεία για να καταλάβετε περίπου τι κάνει ο οργανισμός μας. 88 επισκέψεις ε, στα κράτη-μέλη και σχετικούς οργανισμούς είχαμε στον τομέα της, θαλάσσιας, της ασφάλειας της θάλασσας, 36 εργαστήρια με, με 1.170 συμμετέχοντες από τα κράτη-μέλη, 34 ε, κύκλους κατάρτισης ε, με εμπειρονόμενες από όλες τις χώρες, 14 σκάφη κατά της ρήπανσης ε, με τα οποία συνεργαστήκαμε και πρέπει να σας πω το 2010 ήταν η πρώτη χρονιά που δεν είχαμε κανένα σχόλιο από το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει ότι η ΕΜΣΑ είναι ένα οργανισμό που βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να σα ευχαριστήσω εκ νέου, να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο και την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου για τι πολύ σημαντικέ σα συνεισφορά, τα σχόλιά σα, τι παρατηρήσει σα, θα τα λάβουμε όλα υπόψη ώστε να βελτιώσουμε το έργο μα και να έχουμε ασφαλέστερε και καθαρότερε θάλασσες που είναι και ο στόχο μα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τομασίνη για τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε. Τόσες πολλές πληροφορίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εν ώψη και του βαβελμένου της ημερησίας μας για σήμερα το απόγευμα, θα έλεγα να περάσουμε αμέσως στη συζήτηση. Αν ξεκολουθούν να υπάρχουν ερωτήσεις, θα μπορούσε να απαντήσει ίσως και το ηλεκτρικό συνέδριο. Αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την συζήτηση. Καταρχήν η συγγήτρια, η κυρία Μακοβάη έχει το λόγο. Και μετά η κυρία Ιβάνοβα. Παρακαλώ κυρία Μακοβάη. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για κάθε μία από τις υπηρεσίες αυτές. Και Maritime Safety Agency Καταρχήν, το οικονομικό του 2010 χαρακτηρίζεται από πολλές ενδυναμίες. Ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές, το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες ε, δημοσίων αγορών. Και αυτό θα ήθελα να υποβάλω συγκεκριμένε ερωτήσεις. Καταρχήν, για τις αγορές. Οι ερωτήσει μου αυτές είναι για πώ ΕΣΑ. Πώς εξασφαλίζονται η σωστή μεταφορά των στοιχείων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πώς εξασφαλίζει η υπηρεσία, ο οργανισμός αυτός να είναι τα στοιχεία σωστά για τις δημόσιες αυτές αγορές. Δεύτερον, πώς εξασφαλίζεται την έγκαιρη πληρωμή, την έγκαιρη εκτελέση των πληρωμών. Τώρα, για το ανθρώπινο δυναμικό. Αναφερθήκατε στον ε, υπεύθυνο για τις ε, ε, εξουσιοδοτήσεις. Δώσατε την εντύπωση ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω. Είναι επισυμβάση ακόμα. Ποιος τον αξιολογεί, πώς ορίζονται οι αρμοδιότητες τους. Αν μου δίνετε απαντήσεις στις δύο αυτές ερωτήσεις, θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων. Τώρα, όσον αφορά την απόδοση πέρσι ζητήσαμε να ζητά ο οργανισμός ε, συγκεκριμένα διαγράμματα για να παρουσιάζει τις αρμοδιότητες αυτές. Τώρα είδαμε ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της ζωής ε, του αποτελέσματος και των ε, διοικητικών διαδικασιών. Πώς εντάσσονται όλα αυτά στο λειτουργικό πρόγραμμα της ΕΜΣΑ, πώς θα τα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον. Αυτά ήταν ερωτήσει προ την ΕΜΣΑ. Τώρα έχω και κάποιε ερωτήσει για τον ΕΑΣΑ. Uh, Οπωσδήποτε θα χαιρόμουν να έχω σαφείς ε, απαντήσεις σε σαφεί ερωτήσει Πάλι όσον αφορά τι ε, δημόσιε προμήθειες. Ποια είναι τα ποσά για κάθε μία από τις ε, δύο μεγάλες Διαδικασίε ε, προμήθεια για τι οποίε ε, το ηλεκτρικό συνέδριο βρήκε να υπάρχουν προβλήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι αυτά τα προβλήματα, με ποιον είναι τα προβλήματα και ποια είναι τα ποσά για τα οποία συζητάμε. Κατόπιν, πώς εξασφαλίζει η υπηρεσία την αδιαφάνεια της διαδικασίας αυτής ε, προμήθειας και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης. είναι δυναμικό τώρα. Πώς εξαφαρίζεται, εξασφαλίζεται την πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες προσλήψεων. Um, and... The point is that, the representatives of the agencies are... Κοιτάξτε, το κυριότερο είναι ότι να ακούνε οι εκπρόσωποι των οργανισμών προσεκτικά για να μας δώσουν τις απαντήσεις μετά. Λοιπόν, οι στις ερωτήσεις για τον Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας. Θα ήθελα να ξέρω πώς εξασφαλίζει η, η οργανισμός αυτός επαρκή τεκμηρίωση της διαδικασίας εποπτείας και πώς εξασφαλίζει την σωστή καταγραφή και συνοχή που δίζεται στα αποτελέσματά της. Και τελευταία ερώτηση. Είχα ήδη μια ανταλλαγή επιστολών με τον ε, διευθυντή του ΕΑΣΑ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμα όσον αφορά τον τομέα ε, σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί ξέρω ότι εκεί υπάρχουν πολλοί από τους βιομηχανικούς ε, κύκλους, γιατί αυτοί είναι οι εμπειρογνώμοντες. Αλλά θα ήθελα τώρα να ξέρω εάν αυτοί οι άνθρωποι πιστοποιούν αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τις εταιρείε από τις οποίες προέρχονται. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Έχετε τέτοιες καταστάσεις. Έχετε να μου πείτε κάτι από αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Μακόβα είναι πολύ... είναι η μας και έχει πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Τώρα η άλλη, κυρία Ιβάνοβα πρώτη. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Μακοβέ για τις προσπάθειές της, έξοχη δουλειά της. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Θαλασσίων Μεταφορών. Ακούσαμε όλοι την, το πρόσφατο ατύχημα με το κουραζιερόπλιο που έδειξε για ακόμη φορά ότι χρειάζεται ετοιμότητα όσον αφορά τα ατυχήματα, ταχεία αντίδραση, διαθεσιμότητα προσωπικού και εξοπλισμού, δυνατότητα βοήθειας γρήγορη σε περίπτωση ατυχήματο και αντιμετώπιση πετρελοκυλίδων εγκαίρως. Σύμφωνα με την ΕΜΣΑ, πάνω από ένα τρίτο του προπολογισμού τη υπηρεσία δαπανάται για την προετοιμασία καταπολέμηση λίδων. Πρώτη ερώτηση. Πώς αξιολογείται η αντίδραση της ΕΜΣΑ όσον αφορά το πρόσφατο ατύχημα κοντά στις Ιταλικές ακτές. Δεύτερον, πώς αξιολογείται τη γενική αποτελεσματικότητα του συστήματος όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης δοθεί θετική αξιολόγηση του ενεκτικού συνεδρίου. Εξακολουθείτε όμω να πιστεύετε ότι υπάρχουν τομεί που χρήζουν βελτιώσεων. Αν όχι, ε, θεωρείτε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ακούσαμε ότι έχετε θετικέ εντυπωσει. παρόλα αυτά υπάρχει κάτι που μπορεί να βελτιωθεί. Ευχαριστώ κυρία Ιβάνοβα. Ο κύριος Καγιάν είναι επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη από διότι ο κ. Χέρτσοκ, ο σκιώδης συγγητής, είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, η κυρία Χέρτσοκ μάλλον, στην Ουγγαρία και μου ζήτησε να υποβάλω εγώ δύο ερωτήσεις προς τους ε, οργανισμούς εκ μέρους της. Και εγώ πρέπει να φύγω αρκετά σύντομα και δεν ξέρω και επειδή έφτασα και καθυστερημένος κατά πόσο αυτά που θέλω να καλύψω έχουν ήδη αναφερθεί. Στρεφόμενος προς το ελεκτικό συνέδριο. Διεξάγονται ανταλλαγέ απόψεων με το ελεκτικό συνέδριο και με τον πρόεδρο, τον κύριο Καλτέρα. Ο κύριο Καλτέρα μας είπε ότι θεωρεί ότι στις υπηρεσίες αυτές υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου ποιες είναι οι εντυπώσεις του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με το πώς, ποιοι είναι οι κίνδυνοι όσον αφορά τον προπολογισμό των υπηρεσιών. Και θα ζητήσω και εγώ, όπως κυρία Μακοβέη, ε, την έκθεση για τη βαθμολόγηση. Benchmark study. Ε, σίγουρα θα υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εκπονηθεί η έκθεση. Εξαρτόμαστε πολύ από αυτό όμως και γι' αυτό υποστηρίζω το αίτημα των συναδέλφων.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 Γιατί χρειάζεστε τόσο πολύ χρόνο, ερωτώ το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χρειαστήκατε. Γιατί έπρεπε να περάσουμε από τόσες πολλές εκδοχές του κειμένου μέχρι να φτάσουμε στην τελική. Το ελεκτικό συνέδριο εντόπισε κάποιες αδυναμίες όσον αφορά τη διαφάνεια και τις δημόσιες προμήθειες, κυρίως τη διαφάνεια όσον αφορά τις προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασφαλείας Αεροπορικών Μεταφορών. Εκ μέρου τη κυρίας Χέρτσοκ θέτω το ερώτημα. Ποια ανταπόκριση της Υπηρεσίας Ασφαλείας Αεροπορικών Μεταφορών όσον αφορά τα όσα είπε το Ελεκτικό Συνέδριο και τι γίνεται με την προετοιμασία εξωτερικής πιστοποίησης και τα σχετικά σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου. Τρίτο ερώτημα. Προς την Υπηρεσία Ασφαλείας Θαλασσίων Μεταφορών. και τη Μονάδα Νομικών και Οικονομικών Ζητημάτων πιο συγκεκριμένα. Ποια είναι τα αποτελέσματα των νέων εφαρμογών όσον αφορά την αποδοτικότητα δηλαδή όσον αφορά την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Ευχαριστώ και Γιον. Άλλα σχόλια δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε κατευθείαν στις υπηρεσίες, στους οργανισμούς. Να στραφώ πρώτα προς τον κύριο Γκουντού για να μας δώσει μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, δηλαδή τις ε, αγορές θα αφήσω τον οικονομικό μας διευθυντή να απαντήσει. Yes, uh, uh, related to the uh, procurement process. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προμηθειών για τον οργανισμό, πιστεύω ότι σε σχέση και με το με την έκβαση, δηλαδή με τα όσα γράφει το ελεγκτικό σύνδεσμο στην έκθεσή του, ε, αντιλαμβάνεστε ότι παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και εκτελούμε πάρα πολύ προσεκτικά τι ε, προμήθειε, προμηθειών, βάσει δηλαδή των όσων προβλέπουν οι δημοσιονομικοί κανονισμοί. Επίσης αναφέρουμε ε, τα σχετικά με τα σχέδια προμηθειών στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο συγκεκριμένα. Άρα υπάρχει και πλήρης διαφάνεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των μελών ε, του Διοικητικού Διαχειριστικού Συμβουλίου. Υπήρξε ένα θέμα σε σχέση με δύο ε, διαγωνισμούς και συγκεκριμένα είχαμε ένα διαγωνισμό για υπηρεσίες καθαριότητας, μια σύμβαση λοιπόν που θέλαμε να ανανεώσουμε για τέσσερα χρόνια. Ένα εκατομμύριο είναι ο προπολογισμό αυτή τη σύμβαση. Περίπου 200.000 ευρώ το χρόνο δαπανούμε για τον καθαρισμό των κτίριων του οργανισμού. Έπρεπε να αναθεί η σύμβαση. Η παρατήρηση του Ελεκτικού Συνεδρίου είχε να κάνει με το γεγονό ότι για τον υπολογισμό των διαφορετικών στοιχείων της τιμής είχαμε κάνει μια διάκριση μεταξύ των βασικών υπηρεσιών που θέλαμε να ε, μας προσφέρονται και κάποιων επιπρόσθετων υπηρεσιών. Είχαμε λοιπόν καθορίσει έναν συντελεστή σημασία 75% βασικές υπηρεσίες που είναι υπηρεσίες τις οποίες ε, οι οποίε μάλλον αντιστοιχούν στην καθαριότητα και είχαμε και 25% catering, παροχή καφέ, με καφέ λοιπά. Παρατήρηση του ελεκτρικού συνεδρίου ήταν ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πολλά από αυτά τα ποσοστά ή τέλο πάντων να οικοδομήσουμε, να φτιάξουμε κάποια σενάρια για την τελική σχέση κόστου ωφέλου των υπηρεσιών που έχουμε λάβει, μάλλον των προσφορών που είχαμε λάβει. Τεχνικά είναι λίγο τα, τα πράγματα, τέλο πάντων θα την υπόψη αυτή την υπόδειξη και στους μελλοντικού διαγωνισμού που θα προκύξουμε θα κάνουμε αυτή την ε, ε, κατανομή. Πρέπει να σας πω όμως ότι η έκβαση ήταν πολύ θετική για τον οργανισμό μας ό,τι αφορά τις προσφορές. 30.000 ευρώ περίπου εξοικονομήσαμε στη διάρκεια του πρώτου έτους με τη νέα σύμβαση. Άρα κάναμε οικονομίες. Η δεύτερη περίπτωση τώρα ήταν ένας διαγωνισμός, τεχνική σύμβαση, στον τομέα της αεροπορίας. Η παρατήρηση του ελεκτικού συνεδρίου στην προκειμένη περίπτωση αφορούσε ένα στοιχείο του κόστους, σε μία δέσμη 10 περίπου ε, στοιχείων κόστους, το οποίο δεν πληρούσε ο ετών, ο υποψήφιος. Στο μέλλον θα φροντίσουμε να τα έχει συμπληρώσει, να τα συμπληρώνει σε όλα τα στοιχεία προσφορές τους. Αλλά δεν επηρέασε αυτό την έκβαση τη συγκεκριμένη διαδικασία διαγωνισμού, γιατί μόνο δύο προσφέροντες υπήρχαν. Ο άλλος προσφέρον δεν ήταν επιλέξιμος και γι' αυτό στο τέλος δεν προέκυψε καμία συζήτηση, επιλογή, δεν χρειάστηκε να γίνει επιλογή να ληφθεί κάποια απόφαση, Θα σαφές ποιος ε, θα γινόταν ανάδοχος ε, της σύμβασης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις προσλήψεις και τη διαφάνεια σε θέματα προσλήψεων. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι η διαδικασία προσλήψεων που ακολουθούμε είναι άκρος διαφανής. Η δημοσίευση των ε, κενών θέσεων ε, είναι διαδεδομένη, ευρύτατη. Το προσωπικό μας συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες επιλογής και σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούμε και από ένα εξωτερικό κέντρο εξολόγηση εδώ στις Βρυξέλλες να εξολογήσει του υποψηφίου. Όλα τα στάδια της διαδικασία επιλογής καταγράφονται. Έχουμε τήρηση πλήρων πρακτικών, αναλυτικών πρακτικών. Το 2010 άσκησε μια κριτική το ελεγκτικό συνεδρίο στο γεγονό ότι δεν δημοσιεύαμε και δεν είχαμε εγκρίνει κάποια κατόφλια και σε ό,τι αφορά τη διαλογή, τη φάση της διαλογής, του screening δηλαδή των υποψηφίων και επίσης κατά την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων. Έχουμε τώρα ένα κατόφλι, ε, είναι 50% των βαθμών ε, στη διάρκεια του screening και 65% ελάχιστη βαθμολογία πρέπει να έχει ένας υποψήφιος για να μπει ε, στους ε, φεντρικούς πίνακες. Δεν θέλουμε να είναι οριστικά και πάρα πολύ αυστηρά τα κατόφλια αυτά, διότι κάποιες φορές είναι τόσο, πολλά, ε, τόσο πολλές υποψηφιότητες και αν είχαμε ένα σταθερό κατόφλι ενδεχομένως να χρειαζόταν να κάνουμε συνεντεύξεις ε, με πάρα πολλούς υποψηφίου για μία μόνο θέση. Υπερβολικά πολλού υποψηφίου για μία μόνο θέση. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε τον τελικό αριθμό υποψηφίων ε, που θα παρουσιαστούν για συνέντευξη. Να είναι ένα συλλογικό αριθμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι επιθεωρήσει. Οι επιθεωρήσει γίνονται στα κράτη-μέλη στο όνομα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο σχεδιασμό και το πρόγραμμα των επιθεωρήσεων είναι κάτι το οποίο συζητούμε με την Κομισιόν και αποτελεί τμήμα του προγράμματος εργασίας. Και το εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση εκθέσεων, οι εκθέσει αυτέ αποτελούν ιδιοκτησία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού εργαζόμαστε στο δικό τη όνομα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει να τι δημοσιεύσει, τι εκθέσει αυτέ. Και κυρίω όταν έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Αυτό που κάνουμε εμεί είναι κάνουμε μια στατιστική, τέτοια στατιστική συνολική έκθεση για το σύνολο των ε, επιθεωρήσεων που διενεργήσαμε κατά το προηγούμενο έτο, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη ε, σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, στους διάφορους τομείς. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα ή ε, κάποιο πρόβλημα με τις επιθεωρήσεις αυτές. Όποτε τίθετο το ερώτημα ή μας ζητεί το πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη έκθεση που δεν ήταν διαθέσιμη γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Φυσικά δεν δώσαμε τα στοιχεία, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είμαστε πρόθυμοι να κοινοποιήσουμε τις εκθέσεις. Ό,τι αφορά τώρα τις συγκρούσεις συμφερόντων, πάρα πολύ λεπτό θέμα. Το λαμβάνουμε υπόψη μας με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα. Όπως είπε η κυρία Μακοβάη, πολύ πρόσφατα της απέφθανα μία επιστολή σε σχέση με μία περίπτωση την οποία μας είχε επισημάνει. Θέλω να σας πω ότι οι ομάδες εμπειρογνωμόνων μας σε θέματα πιστοποίησης ε, ε, είναι λίγοι, δεν έχουμε πληθώρα εμπειρογνωμόνων και απευθυνόμαστε στον κλάδο, ε, στα κράτη-μέλη. Επειδή εδώ και 8 χρόνια έχουμε εμεί αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Σε εθνικό επίπεδο, δυστυχώ, ε, σε εθνικέ διοικήσει δηλαδή, δεν υπάρχει επαρκέ προσωπικό στον τομέα αυτό. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να επευθυνθούμε στον κλάδο στη βιομηχανία. Τι κάναμε λοιπόν. Υιοθετήσαμε μια διαδικασία πιστοποίησης άκρος αυστηρή, την οποία επικύρωσε ο Διεθνής Οργανισμός ε, της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, ΔΟΠΑ, Διεθνούς Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και η Federal Aviation Administration. Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται μόνο από ένα άτομο. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά από πάνελ και κάποιες φορές και από όλους ε, τους διευθυντές του οργανισμού. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συλλογική λοιπόν λήψη αποφάσεων μπορεί να καταργηθεί, να εξαλειφθεί οποιοδήποτε κίνδυνος σύγκρουση συμφέροντος από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο, από τη βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκουντού. Ευχαριστούμε για τη σύντομη και περιεκτική απάντηση, τις απαντήσεις σας θα δώσω το λόγο στην ΕΜΣΑ και θα ζητήσω για μια εξίσου σύντομη και περιεκτική απάντηση και από εκείνη την πλευρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Όταν είπα ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, δεν ήθελα να δημιουργήσω την εντύπωση ότι πετύχαμε τον τελικό στόχο. Συνεχίζεται η διαδικασία, πολλά διδάγματα, χρειαζόμαστε πολλά μαθήματα. Υπάρχει μεγάλη προθυμία από την πλευρά μας για συνεχή βελτίωση όσον αφορά τις διαπραγματευτικές διαδικασίες. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, υποβάλλουμε έκθεση μέσω της ετησίσιας εκθέσεως. Σε ειδικό παράρτημα παρέχουμε τις πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά το σχεδιασμό των δημοσίων προμηθειών, αυτό είναι ένα κομμάτι των συζητήσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του προγράμματο εργασιών. Ήδη στο προκατατικό πρόγραμμα εργασιών, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση των δραστηριοτήτων προμηθειών για τον επόμενο χρόνο και στο τελικό πρόγραμμα εργασιών που υθετείται το ε, Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο, υπάρχει συγκεκριμένο παράρτημα που παρατίθενται όλοι σχεδιασμένε όλοι σχεδιασμένες προμήθειες κατά δραστηριότητα, ε, κατά κονδύλι, κατά χρονοδιάγραμμα, κάτι που απαιτεί ο δημοσιονομικός ε, κανονισμός. Τώρα, η εκτέλεση των πληρωμών ε, που το ζήτησε η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου, το εξετάσαν το θέμα Έχουμε ειδικό παράρτημα τώρα στην ετήσια έκθεση για καθυστερήσεις και σεβασμό ε, χρονικών ορίων σε αυτό το θέμα αυτό και έχουμε εισαγάγει και τα εργαλεία παρακολουθήσεως, εποπτείας, μηνία σε εσωτερικό επίπεδο για τη δίκηση. Ξέρουν ποιες αποδείξεις έχουν καθυστερήσει και τιμολόγια και αν υπάρχει κάποια δικαιολογία για την καθυστέρηση, αν χρειάζεται να γίνει κάτι. Τώρα, υπεύθυνο για τα λογιστικά ε, αυτό ήταν σχόλιο της εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου. Πράγματι ο αρμόδιος για τα λογιστικά ήταν ένα, η θέση του ήταν προσωρινή, διευθετήθηκε το θέμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επισήμως διόρισε τον υπεύθυνο για τους λογαριασμούς. Ε, έγινε μια διαδικασία αξιολόγησης. Υιοθετήθηκε η ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο όπου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ρόλο να παίξει στη διαδικασία αξιολόγησης και σαν συνυπογράφων μέλος και, και σαν αρχή ε, υποβολής εφέσεων. Άρα στην αξιολόγηση των λογιστικών στοιχείων ε, που δίνει υπεύθυνο λογιστικά συμμετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, τώρα το διάγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο ψήφισμα για την απαλλαγή. Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο έχει δίνει προστιθέμενη αξία όσον αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες της ε, υπηρεσίας. Η κυρία Ιβάνοβα έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούσαν την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολεμήσεως της Ριπάνσος. Αληθεύει ότι είναι απορροφά τα περισσότερα χρήματα από τον υπολογισμό αυτή η δραστηριότητα. Αληθεύει επίσης ότι έγινε αξιολόγηση, ενδιάμεση αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δείχνει ότι αυτά τα χρήματα όσον αφορά την πρόληψη και την αντίδραση απαιτούνται σαν πόροι, διότι εξασφαλίζεται μια υπηρεσία με προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας δώσω κάποιες ενδείξεις. Η δραστηριότητα, μάλλον η εποπτεία μέσω δορυφόρων για τον έλεγχο υπάρξεως πετρελοκυλίδων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, έγινε διαπραγμάτευση οπότε οι τιμές είναι φθηνότερες για κάθε κράτος μέλος από ό,τι αν είχε διαπραγματευτεί διμερός με την αρμόδια με τις λίγες υπηρεσίες που μπορούν να παράσουν στις υπηρεσίες ε, εικόνων μέσω δορυφόρου. Αν δείτε τα στοιχεία ε, χρησιμεύει σαν αποτρεπτικό μέτρο αυτή η υπηρεσία. Από 1,38 πετρελοκυλίδες αναφωτογραφία που είχαμε το 2008 Πήγαμε στις 0,71 το 2010. Όσον αφορά τα σκάφη, η υπηρεσία ε, αναμονής που χρηματοδοτείται το κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επιτρέπει στα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετο δυναμικό σε περίπτωση ε, μεγάλου ατυχήματος, όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα με, την Κώστα, με το Κώστα Κονκόρδια ε, με σκάφη που δεν θα ήταν διαθέσιμα για τις κυβερνήσεις σκάφη με μεγαλύτερη χωρητικότητα και δυναμικότητα που είναι σε κατάσταση αναμονής. Μετά για την απλούστευση των διαδικασιών υπευλήθη ερώτημα και τι κάνουμε όσον αφορά το σύστημά μας. Χρησιμοποιούμε το ABAC. Αυτό είναι το σύστημά μας της υπηρεσίας και το χρησιμοποιούμε αυτό και σαν τρόπο βελτιώσεως της αναλύσεως των ε, απορρίψεων κάποιων οικονομικών προτάσεων και μαθαίνουμε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις ε, των αρμοδίων επαλλήλων μας και προσπαθούμε να έχουμε κεντρική οργάνωση των αποστολών μέσω του ε, εσωτερικού ελέγχου. Έχουμε εμπειρογνώμους ασχολούνται με την ε, αποζημίωση αποστολών οπότε έχουν μειωθεί απορρίψει απορρίψεις γιατί ακολουθείται σωστή διαδικασία. Αυτά είναι τα μαθήματα που μάθαμε ε, σχετικά με τις ε, δραστηριότητές μας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κυρία Τομασίνη. Ένα ερώτημα είχε απευθυνθεί προς το ελεκτικό συνέδριο θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Γκαλέα να μα δώσει μια συντομότατη απάντηση, διότι μα τελειώνει ο χρόνο. Ο κύριο Γκαλέα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβή ε, για τα σχόλιά τη και τι παρατηρήσει τη. Πρέπει να τονίσω ότι το ελεκτικό συνέδριο εκτιμά το ενεργό τη ενδιαφέρον και τις αποτελεσματικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική, έλεγχο του χρήσεω του ευρωπαϊκού προπολογισμού από τι υπηρεσίε, το ελεκτικό συνέδριο θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ούτω ώστε αποτελεσματικά να υποστηρίζει το έργο τη Επιτροπή σα. Θα ήθελα επίση ευχαριστήσω και του εκπροσώπου των δύο υπηρεσιών, ασφαλεία θαλασσίων μεταφορών και ασφαλεία αεροπορικών μεταφορών, και προσεκλήθη να εκπροσωπήσω το ελεκτικό συνέδριο αντί του κυρίου Οσέ, που είναι αρμόδιος για τους ελέγχου των διαφόρων οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Μου ζήτησαν να διαβιβάσω τη λύπη του, διότι ήταν αναπόφευκτη απουσία του σήμερα, αλλά θα είναι εδώ προσωπικά ο ίδιος ε, στην επόμενη συνεδρίαση όταν θα συζητήσετε την έκθεση του εισηγητού ε, που θα ασχοληθεί με το θέμα των οργανισμών, των υπηρεσιών της Ενώσεως. Τώρα, όσον αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας Μακοβέη και του κυρίου Γκάιερ, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το ελεκτικό συνέδριο δημοσίευσε ειδικέ εκθέσεις για κάθε μία από τις 32 υπηρεσίες. Και στις εκθέσεις αυτές έχει τοποθετηθεί επί της εξοπιστίας των λογιστικών, των υπηρεσιών, νομιμότητας και της ε, ε τακτικότητας των συναλλαγών ε, επί των οποίων βασίζονται τα λογιστικά στοιχεία. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση, ε, ε, συμπεριλάβαμε όταν χρειαζόταν και συμπληρωματικά σχόλια στις περισσότερες εκθέσεις και όχι σε όλες. Τα σχόλια αυτά πρωταρχικά αφορούσαν δημοσιονομικές, ε, δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα. Τα περισσότερα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου σχετιζόταν με το υψηλό επίπεδο των μεταφορών κονδυλίων που μεταφέρθηκαν το 2011. Δεν ξέρω αν η κυρία Μακοβέη κατανόησε αυτού του είδους τις μεταφορές όταν μιλούσε για τις μεταφορές. Αν αναφερόταν σε αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο, των κονδυλίων που μεταφέρονται από το 2011, σημείωσε το ελεκτικό συνέδριο ότι υπήρχαν τέτοιες μεταφορές για εννέα υπηρεσίες και στι ειδικέ εκθέσει συμπεριλαμβάνονται οι κατάλληλε πληροφορίε. Σχολιάσαμε επίση και τι διάφορε αδυναμίε των οργανισμών και των εσωτερικών του συστημάτων ελέγχων, έλλειψη διαφανεία όσον αφορά τι διαδικασίε πρόσληψη, μη συμμόρφωση με τι διαδικασίε προμηθειών, μη συμμόρφωση με του δημοσιονομικού κανονισμού. Τώρα, όσον αφορά το σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε όσον αφορά το αναμενόμενο έγγραφο το οποίο απεκαλεί η έκθεση βαθμολόγησης των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Θα ήθελα να προβώ σε μια διευκρίνηση. Όταν αναφέρεται κανείς στην 17η εκδοχή των λόγων εγγράφου, πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε κάποια παρεξήγηση, πιθανότατα. Η αναφορά ήταν 1,7. 1,7. Ίσως να θεωρήθηκε 17. Όχι εκδοχή 1,7 όπως είναι το σωστό, αλλά 17 ερμηνεύτηκε και αυτό θεωρείται ότι είναι 17η. Ίσως αυτό να βοηθάει και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Να πω κύριε Πρόεδρε ότι συμμερίζομαι την ησυχία και της κυρίας Μακοβέη και του κυρίου Γιάνν Σκάιερ. Ανησυχία όσον αφορά το έργο του ελεκτικού συνεδρίου επί του συγκεκριμένου εγγράφου. Έχουμε δεσμευθεί να έρθουμε στην Επιτροπή με το έγγραφο, το οποίο θα εμπεριέχει τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια εγχειρήματο αξιολογήσεως των υπηρεσιών με βάση το κόστος. Για την ώρα έχουμε οικονομική διαχείριση, επιχειρησιακή αποδοτικότητα, διοικητικό κόστος από πλευρά συγκρίσεων στοιχείων. Δεν έχουμε ακόμα τι αναγκαίε πληροφορίε για να βασίσουμε πάνω σε αυτές μια έκθεση που θα αφορά τη βαθμολόγηση των υπηρεσιών βάσει το κόστος. Οι κανόνες που μας διέπουν και η διαδικασία του ελεκτικού συνεδρίου δεν επιτρέπει να δώσουμε σχέδιο κειμένου. Ο εσωτερικό μας κανονισμό απαιτεί να ακολουθήσουμε τους δικούς μας κανόνες για εφαρμογή και διάφορους άλλους κανόνες των συνθήκων και συνεπώς από τη στιγμή που το ε... θα συνεχίζεται η συζήτηση τώρα και ο Πρόεδρος είπε στην Επιτροπή σας ότι το δεύτερο τριμηνό αυτού του μήνα θα είναι η περίοδος η χρονική κατά την οποία θα υποβληθεί το εγγράφο. Το ελεκτικό συνέδριο έχει αποδείξει ότι προσπαθούμε πάντα να δίνουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να καταλάβει όμως η Επιτροπή ότι μπορούμε να δίνουμε πληροφορίες μόνο όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας και όταν μπορούμε να τι δώσουμε τις πληροφορίες βάσει των δικών μας εργασιών Ω εξωτερικό ελεγκτικός φορέας. Οι περισσότερε πληροφορίε που ίσω να χρειάζεται η Επιτροπή σα πιθανότατα είναι πλέον προσβάσιμοι και διαθέσιμες από τις ίδιες τις υπηρεσίες οι που θέλετε και όχι από πλευράς ελεκτικού συνεδρίου που είναι εξωτερικός ελεκτικός φορέας. Τέλος, όσον αφορά τα σχόλια, το αίτημα του κ. Γκάιγερ για πληροφορίες, θα ήθελα να παραπέμψω στην επιστολή της 18 η Νοεμβρίου του Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπου εκεί ο Πρόεδρος μας τόνισε ότι το ελεκτικό συνέδριο παρατηρεί γενική βελτίωση των επιδόσεων των υπηρεσιών Όπω στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασία και διαβίωσης και ζωής. Είναι βελτιώσει που δεν οφείλονται μόνο στη, στην ιστορική υποβολή εκθέσεων του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά και λόγω της επαγρύπνησης της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, που οδήγησε σε ευαισθητοποίηση μεγαλύτερη στις υπηρεσίες όσον αφορά τους κινδύνους. Και αυτό επηρεάζει θετικά βεβαίως τις επιδόσεις των εν λόγω οργανισμών. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαλία. Έχουμε μόλις 20 λεπτά στη διαθεσή μας για το επόμενο σημείο που έχουμε στην ε, ημερήσια διάταξη. Στις 29 Φεβρουαρίου του 2012 η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα συζητήσει την έκθεση 5 Μαρτίου που Προθεσμία Υποβολή Τροπολογιών, 5 Μαρτίου 2012. Θα έχουμε και άλλη δυνατότητα να συζητήσουμε την έκθεση ε, εις βάθος Οπότε θα έχει το τελικό λόγο πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Μακοβίου. Κύριο Στάις έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έπρεπε να είμαι σε τρεις ε, επιτροπές ταυτόχρονα, κάτι το οποίο μάλλον δεν είναι και τόσο εύκολο. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή. Επικεντρωνόμαστε εδώ στους οργανισμούς. Θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτρια να δει και την ε, έκθεση της προηγούμενης χρονιάς, έγιναν κάποιες αρκετά έντονες παρατηρήσεις για ορισμένους οργανισμούς, ότι υπάρχει δηλαδή σύγκρουση, αντιπαράθεση μεταξύ του προσωπικού στην ΕΦΣΑ παραδείγματος χάρη, κάποια Κάποιοι υπάλληλοι της ΕΦΣΑ πηγαίνουν στην γεωργοδιατροφική βιομηχανία. Το είδαμε πρόσφατα αυτό. Ή οργανισμός φαρμάκων. Αντίστοιχη περίπτωση. Κάποια άτομα έφυγαν από την υπηρεσία αυτή και πήγαν στην φαρμακοβιομηχανία να εργαστούν. και έχουμε ζητήσει κάποιες διευκρινίσεις. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει από τη στιγμή που συζητάμε την απαλλαγή να προσέχουμε τέτοιες περιπτώσεις πιθανής σύγκρουση συμφερόντων. Όταν επαναλαμβάνω έχουμε άτομα τα οποία περνούν από, την, ε, από κάποια υπηρεσία σε ένα κλάδο της βιομηχανίας. Θέλω να δω αν η συγγήτρια θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αλλιώς να υποβάλω εγώ σχετική τροπολογία. Σημαντικό, λέει ο πρόεδρος. Σας δώσω το λόγο στην κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Βεβαίω και είναι ένα από τα βασικά μελήματα που έχω για αυτή την έκθεση. Δηλαδή η σύγκρουση συμφερόντων γιατί επηρεάζει πάρα πολύ και τη δαπάνη των πόρων και πολλά άλλα πράγματα. Μάλιστα προτίθεμαι και έχω ε, προβλέψει να επισκεφθώ ορισμένους οργανισμούς ακριβώς για αυτό το ζήτημα της ε, σύγκρουσης συμφερόντων. Και υπάρχουν και κάποιοι που από τον κλάδο, το συγκεκριμένο, έρχονται παραδείγματο χάρη στην υπηρεσία για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Έξω και επέβαλα ερώτημα στον διευθυντή. Έχουμε και ε, πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν κατάλαβα πολύ καλά από την απάντησή σας. Αν εγώ είμαι μία εμπειρογνώμων από την βιομηχανία και έρχομαι μετά στην ε, υπηρεσία, στον οργανισμό να δουλέψω, μπορώ να πιστοποιήσω αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η βιομηχανία από την οποία προερχόμουν. Δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Πώ μπορούν να πιστοποιούν δηλαδή αεροσκάφη αυτοί που δούλευαν πριν για τι ε, επιχειρήσει αυτέ. Πάντω σα ευχαριστώ για την παρουσία σα σήμερα εδώ. Ίσως μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας όλα αυτά τα οποία μας είπατε προφορικά θα μπορούσαμε να τα είχαμε σε έγγραφη μορφή, σε μια επιστολή, ως follow-up αυτής της ακρόασης. Ακριβώς αυτό που είπατε, δηλαδή αν μπορείτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μας το στείλετε με όλα τα νούμερα, με όλα τα επιχειρήματα. Τέλος για το ελεγκτικό συνέδριο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η έκθεση benchmarking, συγκριτική αξιολόγηση, που έχει να κάνει με διάφορα θέματα διαρθρωτικά για τους οργανισμούς, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και η σύγκρουση συμφερόντων, Υποτίθεται ότι θα ήταν ε, έτοιμη τον Οκτώβριο. Μετά αναβλήθηκε για το Δεκέμβριο. Μετά ο πρόεδρο του Ελληνικού Συνδρομικού Καλντέρα, γιατί έχουν και τα αρχεία, είπε δημοσία ότι. Δεν είναι έτοιμο ακόμη. Δεν είμαστε παιδιά. Έχουμε φτάσει στα μέσα Ιανουαρίου. Και επιμένω ότι πρέπει να μας δοθεί αυτή η έκθεση. Και θα τα λάβω όλα αυτά υπόψη όταν θα συζητήσουμε την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση της ε, συγγετρίας. Να απαντήσετε λέει γραπτά στις ερωτήσεις. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε το σημείο 10. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των διαφορών οργανισμών. Και περνάω στο σημείο 11. Απαλλαγή στις κοινέ επιχειρήσεις για το 2010. Πάλι η συγγήτρια είναι η συνάλφος, κυρία Μακοβαή. Καταρχήν όμως ο πρόσωπος του ηλεκτρικού συνεδρίου έχει το λόγο. Χαιρετίζω επίσης τους ε, εκπροσώπου τη κοινή επιχείρηση πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα, καθώ επίση και την Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για την ΙΤΕΡ και την ανάπτυξη πυρηνική σύνδεξη. Ο πρώτο θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάντισλαβ Μπάλκο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγγήτρια, κύριε Μακοβέη, αγαπητοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω την τρίτη πλέον έκθεση αυτό το διήμερο. Πρόκειται συγκεκριμένα για τον έλεγχο 2010, έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις συμπράξεις ως ε, αναφέρον για, τα, για τα έξι αυτές ε, συμπράξεις κάτω από τις Γενικές Διευθύνσεις RCH και INFSO. Θα σας πω ότι ο Γιώργος Φαζάκας ε, είναι υπεύθυνο για την σύμπραξη ΣΕΖΑΡ υπό την γάμα δέλτα Move. αλλά θα τον εκπροσωπήσω. Η εντολή του συνεδρίου είναι λοιπόν να ερευνήσουμε διάφορα θέματα και σύμφωνα με το 287 άρθρο της Συνθήκης Ατλητικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την ειδική εντολή για την διεξαγωγή του ελέγχου των λογαριασμών των συμπράξεων. Δεύτερον, να ελέγξει την κανονικότητα και την νομιμότητα των υποκείμενων συναλλαγών, όπως αναφέρεται σε ειδικέ ειδικές εκθέσεις για κάθε κοινή επιχείρηση, που σας παρουσιάσω. Τρίτον, έκδοση γνωμοδοτήσεων για τους ε, χρηματοοικονομικούς κανονισμούς, αλλά οποιοδήποτε άλλο ε, θέμα δημοσιονομικής διαχείρισης, εφόσον κληθούμε να κάνουμε μια τέτοια αναφορά. Επίσης, ε, είχαμε για να σας αναφέρω την έκδοση της γνωμοδότησης 4-2008 για την, τον οικονομικό κανονισμό της σύνδεξης, για την κοινή επιχείρηση ενέργειας, την γνωμοδότηση 2 του 2010 για τους χρηματοοικονομικούς εικόνες του ΣΕΖΑΡ και του 2 του 2011 για τους χρηματοοικονομικούς κανόνες της κοινή επιχείρησης ε, καθαρή ουρανή. Και τέταρτη ε, αρμοδιότητα, διεξαγωγή ελέγχων για την ε, χρηστή οικονομική διαχείριση, τους λεγόμενους ελέγχους επιδόσεων που αναφέρονται και στις ειδικέ εκθέσεις. Σε ό,τι αφορά τι ειδικέ ε, ετήσιε εκθέσει, ξεκινήσαμε την εργασία μα πάνω στη νέα γενιά κοινών επιχειρήσεων τον Απρίλιο του 2008. Τότε δύο μόνο ήταν επιχειρησιακέ, ε, η Fusion for Energy και το Caesar. Και εκδώσαμε ειδικέ ε, ετήσιες εκθέσει για αυτέ τι δύο κοινέ επιχειρήσει. Το 2009 Είχαμε άλλε τρει επιχειρησιακέ επιχειρήσει, ε, το ΙΜΗ, Clean Sky, καθαρό ουρανή δηλαδή, και Artem. Και άλλε δύο ε, το 2010, Ένια και FCH. Ε. Έχουμε εκδώσει λοιπόν τις αντίστοιχες εκθέσεις. Στόχος και το 2010 ήταν με τις γνωμοδοτήσεις μας να εκφράσουμε την άποψή μας για την αξιοπιστία των λογαριασμών καθώς και για την κανονικότητα και νομιμότητα των συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά ε, το ΙΜΗ, το Fusion for Energy και όλες τις άλλες κοινέ επιχειρήσεις, θα δείτε τις ε, ε, απόψεις μας. Είχαμε αιτιολογημένη γνώμη όμως μόνο για το ΕΝΙΑΚ σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το θέμα που προέκυψε με την παρουσίαση της υλοποίηση ε, των, των προϋπολογισμών. Σε ό,τι αφορά τώρα την κανονικότητα και την νομιμότητα, εκεί ήταν σαφής, ξεκάθαρη απόψή μας, δηλαδή κανένα πρόβλημα για όλους τους για όλες τις κοινοπραξίες. Θα ήθελα τώρα να πω ότι ήταν σχετικά χαμηλή, ε, χαμηλά τα ποσοστά υλοποίηση. Υπήρχαν καθυστερήσεις για την εφαρμογή κάποιων δραστηριοτήτων, για την υλοποίηση, τη λειτουργία των, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, επικύρωση των συστημάτων κτλ. Τώρα, είπαμε ότι δεν υπήρξε εκμετάλλευση των χρηματοοικονομικών πόρων. Το σχέδιο άργησε να επικυρωθεί, να επικυρωθεί. Εξίσου αργά ξεκίνησε και η πρόσκληση υποβολή προσφορών σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. ...98 εκατομμύρια ευρώ πέρασαν στις δεσμεύσεις υποχρεώσεων το 2010 και είχαμε και 64 εκατομμύρια κύρωση πιστώσεων πληρωμών. Αυτά όλα που λέω αφορούν το ίμι. Παρ' όλα αυτά εκεί είχαμε πρόοδο σε κάποιες άλλες πτυχές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις 14 Δεκεμβρίου του 10 εγκρίθηκε η εξπόστη στρατηγική για την αξιολόγηση της νομότητας και κανονικότητας των υποκειμένων συναλλαγών. Θα δει το συνέδριο ε, το αποτέλεσμα των εσωτερικών αυτών ελέγχων στο πλαίσιο του ελέγχου του 2011. Όπως και για τις περισσότερες κοινέ επιχειρήσεις κάνουμε σχόλια για τις ε, συμφωνίες τις διάφορες που έχουν επιτευχθεί και στο Fusion for Energy και στο ΙΜΗ. Για το ΙΜΗ έχουμε να πούμε ότι τη συμφωνία αυτή δεν είχε συναυθεί. Το ίδιο σημαίνει και με το Fusion for Energy οι μόνιμες εγκαταστάσεις δεν έχουν διατεθεί για την κοινή επιχείρηση αυτή όπως προβλεπόταν. Σε σχετική συμφωνία όλες οι κοινέ επιχειρήσεις έχουν να κάνουν και με το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή της Επιτροπής και με τον κύριο Φαζάκας και με το προσωπικό. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό. Είχα την ευκαιρία να το συζητήσω και με τον Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας στερικού Ελέγχου το Σεπτέμβριο του 2011 με τον κύριο Γκρέι και στις τρεις γνωμοδοτήσεις σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς κανόνες των ε, κοινών επιχειρήσεων αλλά και επανειλημμένα στις ετήσιες ειδικέ εκθέσεις για τις κοινέ επιχειρήσεις ε, το συνέδριο αναφέρεται στο άρθρο 71 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού του κανονισμού 2433 του 2002. κανονισμό 2343 του 2002. με βάση το οποίο ο εσωτερικό ελεγκτή επιτροπή έχει τι ίδιε εξουσίε σε σχέση με του οργανισμού, άρα και με τι κοινέ επιχειρήσει, ό,τι αφορά τα τμήματα τη Κομισιόν. Χαίρομαι που χάρη και στις προσπάθειες ε, του συνεδρίου έχει επιτευχθεί πρώτα σε σχέση με την διευκρίνηση αυτού του ζητήματος και τώρα όλες οι κοινέ επιχειρήσεις δέχονται το ρόλο του ελληνικού ε, συνεδρίου. Ένα θετικό παράδειγμα σε ό,τι αφορά το Fusion for Energy λάβαμε κάποιες ε, από τις τροποποιήσεις που θα κάνουν στο δημοσιονομικό τους κανονισμό. Είχαμε κάνει 50 παρατηρήσεις, δέχτηκαν τις 48. Πολύ επικοδομητική προσέγγιση. Και δείχνει ότι επηρεάζει το συνέδριο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Fusion for Energy ενέκρινε τις τροποποιήσεις αυτές ε, στο δημοσιονομικό κανονισμό θα συνεδρίασε στις 24 και 25 Νοεμβρίου του 2011. Για το Fusion for Energy να μιλήσω ακόμη λίγο και να πω ότι πρέπει να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τη φάση κατασκευής του ΙΤΕΡ. Έχουμε επανειλημμένο στον ετήσιας ειδικέ εκθέσεις και στην έκθεση του 10 ε, το θέμα αυτό και με σημειώνω με ικανοποίηση ότι τελικά λύθηκε το θέμα μετά από το συμβασμό Συμβουλίου Κοινοβουλίου και Κομισιόν στις αρχές Δεκεμβρίου του 2011. Το συνέδριο θα παρακολουθήσει και στη συνέχεια πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως ε, έχετε καταλάβει από τη μέχρι τώρα παρουσίασή μου, ένα πάρα πολύ σημαντικό επίκαιρο θέμα αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις. Δεν ε, έχουν να κάνουν μόνο με προβλήματα ή προκλήσεις, αλλά βλέπουμε να υπάρχουν και συνέχεια εξελίξεις. Επομένως, έτσι μόνο και μόνο για ε, να σας δώσω δύο παραδείγματα και για να σας ενημερώσω θα επιστήσω την προσοχή σας σε δύο ε, συγκεκριμένες ε, σκέψεις στην πρόταση της Κομισιόν για μία απόφαση του Συμβουλίου που αφορά το ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος Ορίζοντας 2020, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020. Στι 30 Νοεμβρίου 2011 παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα η Κομισιόν. Στο τέταρτο εδάφιο του πρώτου παραρτήματος, εκεί η Κομισιόν θέτει το ενδεχόμενο να συνδυαστούν ένιακ και άρτεμις σε μία πρωτοβουλία. Και στα σχόλια μετά το σημείο 7 ε, του Legislative Financial Statement αναφέρει τη δυνατότητα να υπάρξουν και νέες κοινέ επιχειρήσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης των εταιρικών προκλήσεων που είναι μέρος του ορίζον 2020. Κύρια ε, εισηγήτρια, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκλησή σας και για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπαλκό. Θα ήθελα να δώσω μέσα το λόγο στην ε, Διευθύντρια της ΕΜΗ και στη σύνδεξη ε, στο θέμα της ε, σύνδεξης για ενέργεια. Παρακαλώ μην μιλήσετε πέρα των πέντε λεπτών. Member of the Parliament, uh, lady. μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω ε, την ε, πρωτοβουλία για τα φάρμακα που θεωρούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα όραμα, οραματική δημιουργία πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα για να προωθήσουμε έναν τομέα ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη βιομηχανία και για την κοινωνία και τη με την ανθρώπινη υγεία. Simply, based. Η αποστολή μα βασίζεται επί των αποδείξεων ότι οι φαρμακευτικέ εταιρείε από μόνε του δεν είναι αποτελεσματικέ όσον αφορά ε, τα, την παραγωγή καινοτόμων και νέων φαρμάκων και ασφαλών φαρμάκων περιμένουν πολύ ασθενεί. Για να αλλάξει λοιπόν η κατάσταση η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα αλλάζει την προσέγγιση με μεγάλα προγράμματα ευρέα εμβελία με βάση δύο βασικών αρχών. Πρώτα απ' όλα, έρευνα πριν από, το, από τα μέτρα ανταγωνισμού. Έχουμε την, ε, μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες ε, που συνεργάζονται ε, συλλέγουν πόρους ε, και κινητοποιούνται επί συγκεκριμένου ε, στόχου. Αυτή είναι η συνεργασία προ-ανταγωνισμού. Και μετά θέλουμε ανοιχτή καινοτομία. Έχουμε περίπλοκες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε πολλές εταιρείε να συνεργάζονται δεν αρκεί. Θα πρέπει να εδραιωθεί συνεργασία με τέρους εκτός της βιομηχανίας, στα πανεπιστήμια, σε μικρομεσές επιχειρήσεις ε, υπάρχουν αυτοί με τους οποίους μας συνεργάζονται, με οργανώσεις ασθενών. Επί πολύ μακρόν η φωνή των ασθενών απουσίαζε από την διαδικασία ανάπτυξη από το φαρμάκων και συμμετοχή ρυθμιστικών φορέων. Αυτά τα κονσόρτσια για να λειτουργούν αποτελεσματικά πρέπει να υπάρχει μια βάση ουδέτερη, αυτόνομη. Uh, για πολλούς λόγους, ούτως ώστε να υπάρχει σωστή, ε, σωστός επιμερισμός της γνώσης και διάδοση σωστή και να υπάρχει και οθή διαχείριση των δημοσίων ε, πόρων ε, στη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Δεν έχω χρόνο να σας πω ότι μόνο μετά από δύο χρόνια επιχειρήσεων ε, τα κονσόρσια μας έδωσαν πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε σημαντικούς τομείς όπως πνευματικές διαταραχές όπως είναι η σχιζοφρένεια, ο διαβήτης, ε, ασθένειες των πνευμόνων και πολύ συχνά τα προγράμματα βασίζονται ε, επί αναφορών των ασθενών στον αφορά τη δράση των φαρμάκων και κινηθήκαμε επίσης και στον τομέα της ασφαλείας των φαρμάκων και πιστεύουμε ότι αναμένουμε και άλλα αποτελέσματα. Για να κλείσω θα πω ότι η βάση των πρώτων επιταγμάτων η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα θεωρείται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα θεωρείται σαν ένα πρότυπο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης καινοτόμων και ασφαλών θεραπείων προφανώς προς, ε, που αυτά θα είναι προς όφελος των ασθενών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκόλμαν για την εκθέση σας. Παρακαλώ, ο κύριος Ρίσκ έχει το λόγο τώρα. So, thank you, Mr. President, and... Uh, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα την εφορή και την πρόοδο ιδρύθηκε με ένα συγκεκριμένο στόχο πριν από 10 χρόνια δηλαδή να παίξει τον ευρωπαϊκό ρόλο σε ένα μεγάλο σχέδιο διεθνές, δηλαδή η ανάπτυξη της, ε, του μηχανισμού ITER σε ένα διεθνές σχέδιο στη Γαλλία. Είναι το επόμενο στάδιο που θα αποδείξει την ε, ε, δυνατότητα πραγματικά πραγματοποίησης ε, της σύνδεξης για λόγους ε, παραγωγής ενέργειας. έχει ένα τεράστιο σχέδιο, ψηλότητα της τεχνολογίας, υψηλότητα του κόστους επίσης και γίνεται σε διεθνές περιβάλλον με έξι άλλους εταίρους. Αμερική, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία και Νότιο Κορέα. Η Ευρώπη έχει το 45% του συνόλου των εργασιών αυτών. Ορισμένα μέλη τη Επιτροπή σα ενδιαφέρθηκαν για το σχέδιο Φιόιτερ και μάλιστα έγινε και μια επίσκεψη στο Κανταράσ στη Γαλλία πέρσι τον Μάη και νομίζω ότι κατόπιν αυτού είσαστε πολύ καλά ενήμεροι για το σχέδιο και την πρόοδό του. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω ορισμένα λεπτά στην ε, ενημέρωσή σας. Όσον αφορά αυτή αυτή την εργασία, από πέρσι τον Μάη επιτεύχθη καλή πρόοδος εκεί επί τόπου. Οι κύριες εξκαφές ολοκληρώθηκαν. Τα πρώτα δύο κτίρια θα ολοκληρωθούν τους τρεις με τέσσερις επόμενους μήνες. Εν τω μεταξύ αρχίσαμε τους διαγωνισμούς για περαιτέρω κτίρια. Ε, χρειάζεται να δώσουμε συνολικά 30 κτίρια και το πιο μεγάλο κτίριο που είναι για το μηχάνημα είναι σε αντικείμενο διαγωνισμού εδώ και 12 μήνες και ελπίζουμε να δώσουμε την σύμβαση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Εκτός από τα κτίρια θα πρέπει να δώσουμε τα περισσότερα ε, εξαρτήματα για την κατασκευή της μηχανής αυτής Υπάρχουν βέβαια κάποια καθυστερήσεις στη Γαλλία και εκτός Γαλλίας, αλλά αυτό είναι σύνηθε σε ένα τέτοιο είδου σχέδιο. Όσον αφορά το πιο σημαντικό ε, στοιχείο, τους τις ε, μαγνήτες, υπάρχει η πρόοδος, υπάρχουν ήδη κατασκευές πρωτοτύπων, ε, επιτυχής κατασκευές και θα αρχίσουμε τώρα την σειρά παραγωγή των ε, των ποινίων αυτών. Προσπαθούμε επίσης να κάνουμε κάποιες ε, βελτιώσεις στην οργάνωση του εφορεί, κάτι που το είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με την αύξηση του προϋπολογισμού μας. Και θα ήθελα να σας πω και εκεί δύο λόγια, που ίσως να ενδιαφέρουν και το Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα μας ζητήθηκε να περιορίσουμε το κόστος του σχεδίου, να μην ξεπεράσουμε δηλαδή τα 6,6 δις ευρώ που είχαν καθοριστεί για το σύνολο της κατασκευής. Μέχρι στιγμής η εικόνα είναι πολύ καλή. Αυτή η εκτίμηση γίνεται γίνει πριν από δύο χρόνια και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να αντιταχθούμε σε μια σειρά αυξήσεων γιατί υπήρχαν και ανάλογες εξοικονομήσεις. Βέβαια η εικόνα αλλάζει με την παρόδο του χρόνου και δεν μπορεί να προβλέψει καλά το μέλλον. Αλλά για δύο χρόνια η απόδοση μας ήταν πολύ καλή. Όσον αφορά την δομή του εφορίν έγιναν σημαντικές αλλαγές που είχαν κυρίως σαν στόχο μία δομή που προσανατολίζεται περισσότερο στο σχέδιο αυτό και ένα νέο ανώτατο διοικητικό προσωπικό τον επόμενο μήνα θα οριστούν οι ε, επικεφαλής του σχεδίου, οι διάφοροι μάνατζερ. Μέχρι στιγμής είχαμε μονάχα κάποιους ε, επισυμβάσει αν θέλετε. Τώρα κάνουμε όμως διάφορες ε, συνομιλίες και θα ελπίζουμε τον επόμενο μήνα να έχουμε τους οριστικούς ορισμούς. Το ίδιο όσον αφορά το διαδικαστικό Προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε ένα έγγραφο όσον αφορά στι εσωτερικέ διαδικασίε τη οργάνωση. Ε, κάποια διοικητικά εγχειρίδια προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή και περιμένουν να τα εγκρίνω. Όσον αφορά τη διαχείριση του σχεδίου αυτού καθεαυτού, που είναι το θέμα που μου απασχολεί περισσότερο, η κατάσταση είναι κάπως πιο δύσκολη. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώσαμε το σχεδιασμό ενός νέου συστήματος συμβατού με ε, κεντρική οργάνωση της Ίντρας, το Καντεράς και με τους άλλους διεθνείς μας εταίρους. Και ε, αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε. Θα έλεγα ότι ίσως απέχουμε ακόμα έξι μήνες περίπου μέχρι να εγκαθιδερθεί οριστικά. Τέλος, σε σχέση με την ανεξάρτητη αξιολόγηση, έχω να πω ότι επιτέχθηκε σημαντική πρόοδος. Πάντα θέλαμε να έχουμε εσωτερικούς ε, ελέγχους. Αυτό το σύστημα εδώ και 18 μήνες είναι πια λειτουργικό. Το αναφέρει το ηλεκτρικό συνέδριο. Πρόσφατα δεχθήκαμε τον ρόλο της εσωτερικής υπηρεσίας ελέγχου της Κομισιόν που συνεργάζονται τώρα με τη δική μας ε, μονάδα για εσωτερικούς ε, ελέγχους συμφωνούν ένα κοινό πρόγραμμα Έχουμε αυτή την ε, Επιτροπή Ελέγχων που είναι υπόλογη στο Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης έχει ξεκινήσει τώρα η ε, πρώτη αξιολόγηση της εφορή ως οργάνωσης στο σύνολό τη. Του των εχθέντων ε, νομίζω ότι προχωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Η κυρία Μακοβέ έχει το λόγο. Thank you, President. Um... I have questions for each of the joint Έχω ερώτηση για τον καθέναν από τους εκπροσώπους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για την ανταλλαγή απόψεων. Να πω για το 2010 χρειαζόμαστε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για αυτές τις ε, συμπράξεις. Πάρα πολλά χρήματα. Χίλια εκατομμύρια ή ένα δισεκατομμύριο. Τώρα σε ερωτήσεις. Είναι πολύ δύσκολο για κάποια κράτη-μέλη να βρουν οικονομικούς πόρους στις αγορές. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να πληρώσουν και επιτόκιο 6% και παραπάνω. Περνάμε από οικονομική στενοπόλη. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Αναφέρομαι στην πρωτοβουλία για τα φάρμακα. Πώς δικαιολογείται ότι στο τέλος του έτους έχετε 71 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα το ίδιο στη σύνδεξη για ενέργεια. 78,8 εκατομμύρια ευρώ είναι το αντίστοιχο ποσό. Και ποιο είναι το επιτόκιο που παίρνει κάθε υπηρεσία από τα ποσά που έχει στην τράπεζα. Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα τώρα. Πώς εξηγείται η χαμηλή χρήση των της αναλήψεως των υποχρεώσεων 6% και των πληρωμών 35% δεσμεύσεις για πληρωμές. Άλλη ερώτηση για την πρωτοβουλία για τον τόμα φάρμακα. Στην ετήσια 6 του 2010 για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων είδαμε ότι η υπηρεσία ασχολήθηκε με την έκθεση την ετήσια της σύμπραξης. Είναι σωστό? Αυτή η υπηρεσία ε, ε, συντάσσει την τελική έκθεση. Γιατί, ποια είναι η προστιθεμένη αξία. Για τη σύμπραξη τώρα, για τη σύνδεξη. Μάρτιο του 2008 ξεκίνησαν οι εργασίες σας. Κινηθήκατε αυτόνομα. Η νέα οργανωτική ξεκίνησε η του 2012 και τα συστήματα για τον έλεγχο των στοιχείων δεν λειτουργούν πλήρω και δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα πλήρω. Πόσο χρόνο χρειάζεστε, Εξάμεινο και γι' αυτό το μηχανισμό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Θα ήθελα και από και των δύο συμπράξεων να λάβω γραπτός μέχρι το τέλος της εβδομάδος αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ. Ja, äh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Συγγετρία, κυρία Μακοβάη. Θα ήθελα πραγματικά και εγώ να υποστηρίξω αυτή την πρόταση της συζητήτριας. Να απαντήσετε σα σύντομα και μετά να έχουμε μια πιο αναλυτική απάντηση γραπτά, παρακαλώ. Δύο συνάδελφοι έχουν ζήσει το λόγο με συμπληρωματικέ ερωτήσει ή τοποθετήσει. Ο Σνόφο Ρούμπιχ πρώτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει για την ΕΤΑΡ. Υπήρξε μακροπρόθεσμος ε, οικονομικός προγραμματισμός που είχε γίνει δεκτός και από τους έξι εταίρους μας. Αυτό νομίζω ότι είχε γίνει όμως σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η ε, πιστοτική κρίση δεν ήταν τόσο έντονη όσο είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα υπάρχουν νέες απαιτήσεις. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Και το ελεκτικό συνέδριο τώρα πώς αξιολογεί την κατανομή του κόστους μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι εταίρων. Αυτή η συμφωνία που πετύχαμε ε, οδηγεί σε μια κατανομή που είναι σύμφωνη με τις ανάγκες ε, του σχεδίου ή θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρώτα ευχαριστώ. Ο συνάδελφος έχει το λόγο. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να αναφερθώ στην Ίτερ μόνο. Και να σας πω τα εξή. Το σύνολο της ε, αντιπροσωπείας ε, των Επιτροπών Προεπολισμού και Ελέγχου Προεπολισμού πήγε στο Καντεράς και ήμουν επικεφαλής και είδαμε πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις εκεί και είχαμε και έκθεση με μια σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων και συστάσεων. Πάνω στις ερωτήσεις αυτές πήρα μια σειρά απαντήσεων προφορικών και ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά θα ήταν καλό η σύσταση που είχαμε διατυπώσει να ξαναεξαστεί από εσά και ίσως να, να τοποθετηθείτε με αυτής και γραπτά. Τι έγινε δηλαδή με αυτές τις συστάσεις που κάναμε μετά την επίσκεψή μας στο Καντερά στο περασμένο Μάη. Ευχαριστώ συναρφιστάς. Γιάννης Κάιερ έχει το λόγο. Ναι, ναι, εντάξει, θα δούμε. Συμφωνήσαμε με την συνάδελφο ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε μία ερώτηση προς τον κύριο Μπρίσκ. Εγώ στο Καντεράς ενημερώθηκα ότι υπήρχαν τεράστια προβλήματα για το, τη σύνδεξη για ενέργεια να υπάρξουν αποθέματα γιατί τα κράτη-μέλη αποσύρουν τα πλεονάσματα που υπήρχαν αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον δεν ξέρω ίσως κάτι δεν ε, κατανόησα σωστά και θα ήθελα να μου το ελέγξετε αυτή τη στιγμή γιατί αυτό δεν είναι σύμφωνο ίσως με τις πληροφορίες της κυρίας Μακοβέη για το πρόγραμμα σύνδεξη για Ενέργεια και τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τις εξοικονομήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σχέδιο ΙΤΕΡ μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν σαν απόθεμα που ίσως θα καλύψει μελλοντικές, ε, μελλοντικές απαιτήσεις ή απορροφώνται ξανά από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κυρία Βολμάιερ. Ε, νομίζω ο κύριος Φρίσκ θα ήταν πολύ ευτυχής αν είχε κάποιο απόθεμα στα χέρια του. Νομίζω δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Έχω μία ερώτηση ε, που ζητήσετε με αυτό το ταξίδι στην, στο Καταράς. Υπήρχαν προβλήματα με τον επαγγελματικό χαρακτήρα των διαγωνισμών προβλήματα δηλαδή με επιχειρήσεις ή με πολύπλοκες ε, μορφές διαγωνισμών κατά πόσον έχει βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου στο οποίο αναφέρει η κυρία πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση πρώτα ευχαριστώ πολύ μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων οι περισσότερες από των οποίων ε, στρέφονται προς τον κύριο Βρίσκο για την ε, σύνδεξη για ενέργεια θα ήθελα να σας παρακολουθήσω να απαντήσετε σύντομα. Ίσως και εσείς όχι παραπάνω από πέντε λεπτά. Και η πολλαπλή ερώτηση που υποβλήθη και θέλω να υποβάλω και εγώ για σας, ε, κατά πόσο μπορείτε δηλαδή γραπτά να απαντήσετε λεπτομερές ε, στις ερωτήσεις της Επιτροπής μας. Κύριε Μπρίξου, σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ. Με τα χαρά να σας δώσω γραπτή απάντηση, όπως μου ζητήσατε. Θα προσπαθήσω όμως και να δώσω τώρα κάποιες προφορικές απαντήσεις. Νομίζω ότι ένα ε, θέμα που εκτέθηκε το ίτερ αφορά το συνέδριο και όχι εμάς. Άρα αυτό δεν το σχολιάζω και έρχομαι στα άλλα θέματα σε ό,τι αφορά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τις εξελίξεις. Σε αυτό το μέτωπο, νομίζω το βασικό σημείο, τουλάχιστον όταν εγώ μπήκα ε, στη δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου, η πρώτη, ε, ο πρώτος έλεγχος ε, έδειξε πάρα πολλά, πολλές συλλήψεις. Και κεντρωθήκαμε τότε σε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε τώρα ένα νέο χρηματοοικονομικό κύκλωμα και ένα προϋπάρχον πρόβλημα που υπήρχε. Έχουμε τώρα κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Υπήρχαν και κάποιες πολύ ε, σοβαρές και θέσεις που έμεναν κενές εκείνη την εποχή του ελέγχου που πλέον από το καλοκαίρι και μετά πληρώθηκαν ε, νέοι τομεάρχες που ανέλαβαν γρήγορα τα καθήκοντά τους και ένα άλλο σχετικό πρόβλημα, τον καιρό τότε που κάναμε τον έλεγχο, η μονάδα οικονομικών και προπολογισμού δεν είχε παρκές ε, προσωπικό. Ολοκληρώθηκε η στελέχωση με τις προσλήψεις και πολλοί οικονομικοί φορείς, απαληθευτές ε, και τα λοιπά έχουν αναλάβει εδώ και κάποιο καιρό τα καθήκοντά τους. Ιδίω λοιπόν σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά κυκλώματα έχουν γίνει πολλά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποθεματικά και την εξοικονόμηση πόρων, αυτό που λέει η κυρία Χολμάγερ είναι σωστά. Όταν ζητήσαμε αύξηση του προπολογισμού, ε, είχαμε ελπίσει να πάρουμε λίγο παραπάνω από τα 6,6 δις ευρώ. Το συμπεφωνημένο νούμερο 6,6 δις δεν περιλαμβάνει έκτακτες ε, προβλέψεις. Γι' αυτό και θέλουμε να φτιάξουμε ένα αποθεματικό για μελλοντικά προβλήματα. Όπως είπα στην προφορική μου παρέμβαση, μέχρι στιγμής έχουν ως εξή τα πράγματα. Κάνουμε σε κάποιες περιπτώσεις εξοικονομήσεις, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυξήσει. Είμαστε πάντως συνολικά σε μια σχεδόν ουδέτερη θα έλεγα θέση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εξοικονομήσεις ε, που κάναμε αντισταθμίστηκαν ε, λόγω της απορρόφησης των αυξήσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους και φιλοδοξίες μου πάντως είναι να προβούμε σε τέτοιες εξοικονομήσεις και στο μέλλον. Γιατί για ένα τέτοιο σχέδιο σίγουρα θα υπάρξουν ε, αστάθμητοι απαράγοντες αρνητικοί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιες θυσίες σε ό,τι αφορά το εύρος του έργου μας. Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος του το έργο αυτό καθορίζεται από τη Συμφωνία ΙΤΕΡ. Άρα πρέπει να παρέχουμε ορισμένα πράγματα, αλλά κάποια άλλα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια περισσότερο. Οπότε εκεί μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένω κάποιες θυσίες και να μείνουμε εντός ε, του προϋπολογισμού των 6,6 δις. Σε ό,τι αφορά τώρα τους συμβατικούς όρους, Πράγματι, έχουμε κάποιες εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε ήδη κάποιους ε, συμβατικούς όρους και κανόνες που αντιληφθήκαμε ότι δεν ανταποκρίνονταν ε, στην αποστολή μας. Έγινε πολύ μεγάλη αλλαγή σε αυτούς τους συμβατικούς όρους πριν από δύο χρόνια και νομίζω ότι αυτό επέφερε κάποιες βελτιώσεις. Οι κανόνες δεν επέτρεπαν σε κάποιες εταιρείε να υποβάλουν υποψηφιότητα, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς. Ενώ εμείς αντιθέτως θέλαμε να διευρύνουμε ε, και να παρέχουμε σε πιο πολλές εταιρείε ευκαιρίε να συνεργαστούμε. Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη τομή. Αυτή τη στιγμή και πάλι εξετάζουμε πώς μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω προσαρμογές σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με ορισμένες, λίγες στον αριθμό, συμβάσεις που είναι σχεδόν στη φάση της ανάθεσης της σύμβασης. Όλα αυτά είναι στο μυαλό μας και είμαστε έτοιμοι να διατυπώσουμε προτάσεις και να εγκρίνουμε τους κανόνες εφόσον το απαιτήσει η κατάσταση της αγοράς. Υπήρξαν και κάποια άλλα ερωτήματα. Το 2010 η υλοποίηση του προπολογισμού δεν ήταν ε, τόσο καλή. Το ΕΦΟΡ ήταν μια νέα οργάνωση τότε. Το 2010 κάποιες από τις πιο μεγάλες συμβάσεις ε, θα συνάπτονταν Εκείνη την εποχή είναι λίγο απρόβλεπτο τι γίνεται όταν ε, γίνονται διαγωνισμοί για την ανάθεση μεγάλων συμβάσεων. Και ανάλογα και με το, το χρονικό ε, όριο, τη, τη, στιγμή του έτους, εξαρτώταν και αν θα υπάρξει αξιοποίηση των πόρων ή όχι. Αυτό και το 2010 δεν ήταν πολύ καλή υλοποίηση. Τώρα, ε, έχουμε μακροπρόθεσμες συνήθως συμβάσεις πενταέτους διάρκειας. Οπότε τότε έχουμε μια σταθεροποίηση. Γιατί έχουμε το σύνολο των πληρωμών από συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί. Άρα έχω ε, πιο πολλές, ε, πιο μεγάλη αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, κοινοβουλευτική επίσκεψη του στο Κανταράς, θα σας απαντήσω αν μου επιτρέπετε εγγράφος. Πολύ ωραία θα ήταν αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας και που μας υποσχεθήκατε επίσης τα γραπτά. Ο κύριος Γκόλμαν για μια πολύ σύντομη απάντηση παρακαλώ. Μάλιστα και εμείς το ίδιο. Θα σας δώσουμε όλες τις απαραίτητες ε, λεπτομέρειες γραπτά. Παρ' αυτά θα ήθελα να σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, για τα φάρμακα. Είμαστε απόλυτα ανεξάρτητα από την υπηρεσία αυτή. Ε, προετοιμάζουμε τις δικές μας εκθέσεις κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το κάναμε και το 2010, θα το κάνουμε και το 2011, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού αυτού για τα φάρμακα. Όσον αφορά τον ισολογισμό μετρητών, ε, είναι σωστά τα στοιχεία που έδωσε η κυρία Βουλευτής ε, για το 2010. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση για το 2011 με ένα περί... αποθηματικό 15,2 ε, εκατομμυρίων. Όσον αφορά την κατανομή του βάρους και την καθυστέρηση του προπολογισμού, είναι σωστό γιατί το 2010 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας μας αυτόνομα και για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε, δημόσιους πόρους αναγκαστήκαμε πρώτα να εξασφαλίσουμε την δέσμευση του ιδιωτικού τομέα και ε, ανακαστήκαμε η διαδικασία να περάσει έτσι κατά το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε λοιπόν ε, αισιοδόξοι ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και μάλιστα ήδη βελτιώνεται. Και όπως θα δείτε στα αριθμικά στοιχεία που θα σας δώσουμε η εκτέλεση του προπολογισμού και όσον αφορά και τις δεσμεύσεις και τις πληρωμές ε, έχει βελτιωθεί σχετικά με το περισμένο έτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πόρτμα, ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας πριν να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Η κυρία Μακουβά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα, Είπατε ότι η δική σας έκθεση. Ε, καλό αυτό. Αλλά για διαβάστε όμως την ετήσια έκθεση το 2010 της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Φάρμακα όπου λέγεται ότι τελειοποίησαν τη δική σας έκθεση. Και θα ήθελα επίσης να ακούσω κάτι από τις δύο κοινέ επιχειρήσεις κοινοπρασίες όσον αφορά το επιτόκιο που εισπράτεται για αυτό το αποθεματικό που έχετε γραπτές πληροφορίες μέχρι τα τέλη της εβδομάδας δεν σημαίνει ότι θα το συζητήσουμε τώρα όταν έχουμε τις λεπτομέρειες. Αν έχετε χρόνο σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα. Όσον αφορά τα επιτόκια. Πρόεδρος διακόπτη. Όχι, για να είμαι ειλικρινής δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Γιατί στις... έχουμε άλλο ένα θέμα σήμερα σε διάταξη που πρέπει να συζητήσουμε και στις 5 έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Πέντε λεπτά έχουμε, δηλαδή, 15 ε, λεπτά έχουμε μόνο, δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε ελεύθεροι βέβαια αν θέλουμε να αλλάξουμε την ημερησία διάταξη. Αλλά πώς είχα καταλάβει θα έχουμε τις γραπτές απαντήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά ένας αριθμός, κύριε Γκόλμαν, έχετε τον αριθμό αυτό να τον δώσετε τώρα, ένα αριθμό. That's possible, but better I think το επιτόκιο πόσο είναι. Εάν όχι, δώστε μας το γραπτό. Καλύτερα. Ωραία. Θα μας το δώσουν γραπτά λοιπόν. Σύμφωνοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γκόλμα, κύριε Μπρίσκο, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις δικές σας παρουσιάσεις. Και κύριε Μπάλκο, θέλετε να πείτε μια πρόταση, ένα λεπτό. Of course, I would θα ήθελα βέβαια να απαντήσω στον κύριο Ρούμπικ. όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συμβολής της Euratom. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι θέμα πολιτικής αξιολόγησης ε, του Κοινοβουλίου και της αρμόδιας υπηρεσίας. Ε. Όσον αφορά για το τι αποφασίστηκε πέρσι το Δεκέμβριο, βέβαια και εκεί τονίζω πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία. Αυτό το κοινοβούλιο με το Συμβούλιο έθεσε κάποια πολιτική συμφωνία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι χαίρομαι ότι η Ρία μπορούσε να βρει αυτά τα συμπληρωματικά χρήματα και έτσι θα μπορέσει να πληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει τον των διεθνών της εταίρων μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας ΙΤΕΡ του 2007. Η κατανομή των τμήματων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων ε, εταίρων, ε, Κίνα, Ιαπωνία κλπ. είναι θέμα διεθνού συμφωνίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που τηρήσετε και το χρόνο που σα είχε δοθεί. Είναι σημαντική αυτή η συζήτηση. Θα την ξανακάνουμε στι 29 Φεβρουαρίου και περιμένω να δούμε τις γραπτές σας ε, απαντήσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Κλείνουμε το σημείο αυτό και χωρίς να χρονοτριβήσουμε περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 13. Η εισηγήτρια η Μόνικα Χολμάιερ και εξ ονόματος της, Επιτρο... της Δουλευτικού Συνεδρίου Ράσα Πουτκεργίτε. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο και παρακαλώ να είστε κατά τον σύντομοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Χαίρομαι που σας δίνω τα αποτελέσματα της έκθεσης ε, ε, μας. Ε, η δική έκθεση αυτή είναι ένα τμήμα της γενικής πολιτικής. Η ποιότητα των τροφίμων είναι θέμα που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό αποφάσισε το συνέδριο να κάνει μια, έναν έλεγχο στο τομέα αυτό. Το σχετικό σχέδιο που εισήχθη το 1992 αφορά ένα σύστημα κατανομής, καταγραφής συγγνώμη, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με την γεωγραφική προέλευση. Επίσης αυτό το πρόγραμμα παρέχει μια δυνητική οικονομική δυνατότητα για τους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων και βοηθάει να παραμείνει ο πληθυσμό στην Ήπεθρο. Η συνολική χονδρική αξία των 964, 964 64 ονομασιών που έχουν καταγραφεί στα ε, τέλη του 2010 ήταν περίπου 15 δις ευρώ. Και παίρνουν και κάποια premium ε, αυτά τα προϊόντα κάποια βραβεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τον έλεγχό μα, θέλησαμε να δούμε κατά πόσον η Κομισιόν έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί αποτελεσματικό τρόπο αυτό το πρόγραμμα. Είδαμε, είναι αρκετά ε, ισχυρό το ισχύον σύστημα ελέγχου για να προστατεύσει ονομασίε από ε, λάθο χρήση ή μη εγκεκριμένη χρήση. Είναι ελκυστικό για του παραγωγού. Το αντιλαμβάνονται, το γνωρίζουν οι καταναλωτέ. Και για να λάβουμε τι απαντήσει, επισκεφθήκαμε 8 κράτη-μέλη έξι από τα οποία αντιστοιχούν στο 85 των καταγεγραμμένων προϊόντων. Και τα δύο από αυτά δεν έχουν ξοπίσει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα. Επίσης κάναμε και μία έρευνα και στα 27 κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το σύστημα ελέγχου. Ο έλεγχος μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται διευκρινήσεις στις νομικές διατάξεις. Δεν καθορίζονται ελάχιστε απαιτήσει ώστε οι έλεγχοι να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές προτού τεθούν ε, στο εμπόριο, διατεθούν στο εμπόριο. Οι κανόνες που περιέχει ο επίσημος κανονισμός για τον έλεγχο τροφίμων και ζωοτροφών είτε είναι πάρα πολύ γενικόλογοι είτε δεν ε, έχουν να κάνουν αυτό το σχήμα, ε, το πρόγραμμα. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαροι οι κανόνες που θα πρέπει να γίνουν για να ανοιχτευτεί αν υπάρχει κακή χρήση ενό προστατευμένη ονομασία. Ούτε τα κράτη-μέλη κάνουν, τα περισσότερα τουλάχιστον, τακτικού ελέγχου. Άρα έχουμε μεγάλο κίνδυνο να μην ανακαλύψουμε τέτοιου είδου ε, κακή χρήση. Και δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο η Κομισιόν πάνω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την ελκυστικότητα του προγράμματο αυτού για του παραγωγού, οι μισέ αρχέ των κρατών θεωρούν ότι ε, είναι χαμηλή η ελκυστικότητα και γιατί είναι η διαδικασία καταχώρησης μακροχρόνια και χρονοβόρα και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα το κατά πόσον ε, οι καταναλωτές γνωρίζουν αυτό το πρόγραμμα, με την ανεξάρτητη έρευνα δίδαμε ότι υπάρχει πολύ χαμηλό ποσοστό αναγνώριση και του λογοτύπου και της όλης έννοιας από τους Ευρωπαίους πολίτες, παρότι σχεδόν και 20 χρόνια τουλάχιστον. Επίσης έγινε η έρευνα αυτή το 2008, δηλαδή προτού γίνει υποχρεωτική η χρήση του λογοτύπου. Δεν βλέπω όμως να έχει αλλάξει η κατάσταση από τότε σημαντικά. Δεν έχει στρατηγική, η Κομισιόν κάποια σαφή στρατηγική για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο πρόγραμμα αυτό. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει στι νομικέ διατάξει να καθορίζονται ελάχιστε απαιτήσει για του ελέγχου των προδιαγραφών των προϊόντων. Μεταξύ των οποίων τι πρέπει να καλύπτουν οι έλεγχοι αυτοί και πόσο συχνά θα πρέπει να διενεργούνται. Θα πρέπει επίση να διευκρινιστεί και το πεδίο τη εφαρμογή το εύρο των τακτικών ελέγχων για να ανοιχνευτεί η κακή χρήση προστατευόμενων ονομασιών. Θα ήθελα επίση να δώσω έμφαση στο γεγονό ότι οι συστάσει αυτέ δεν ε, θα πρέπει να δημιουργήσουν ε, τη δημιουργία περαιτέρω στρωμάτων ελέγχου ή μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Δεν ζητούμε δηλαδή περισσότερους ελέγχους, αλλά καλύτερους ελέγχους ως ελεγκτικό συνέδριο. Η μεγαλυτερη γραφειοκρατια δεν ζητουμε δηλαδη περισσοτερου ελεγχου αλλα καλυτερου ελεγχου ω ελεγκτικο συνεδριο η ευρωπαικη επιτροπη θα πρέπει επίση να συμπεριλάβει ε, και τους ελέγχους των κρατών μελών ε, στο σχέδιο των τακτικών ελέγχων που διενεργεί στα κράτη-μέλη. Και τέλος, θα πρέπει να αναπτύξει η Κομισιόν μια στρατηγική για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ευαισθητοποίησης και ε, γνώση για αυτό το πρόγραμμα και να βρει πιο αποτελεσματικού τρόπου για να το προωθήσει. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουμπερτούκη, για την έκθεσή σα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην ε, συνάδελφο Μόνικα Χόλμα, την εισηγήτριά μας. Äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω καρδιότατα την ε, κυρία Μπουτπεργκίτε για τη θαυμάσια συνεργασία και για την συνεχή της διαθεσιμότητα να μας δίνει απαντήσεις και επίσης για την ανάλυση που μας έκανε και την γενική της πρόθεση να μας ανοίξει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πλήρως την εργασία του ηλεκτρικού συνεδρίου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν, η οποία κατόπιν θέλησε να συζητήσει αναλυτικά τα προβλήματα μαζί μας. Είχαμε λοιπόν πάρα πολύ έντονες συζητήσεις για το θέμα. Συμμερίζομαι την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου που αφορά το πόσο γνωστές είναι αυτές οι ονομασίες προέλευσης και θα πρέπει να φροντίσουμε αυτές οι δύο ονομασίες ε, προέλευσης να γίνουν πολύ καλύτερα γνωστές. Επίσης, ε, απέκτησα κάποιες εμπειρίες ότι αν κάποιος παρόλο το screening θεωρεί ότι θέλει να δηλώσει ένα τέτοιο προϊόν με ονομασία προελεύσεως ε, πρέπει να διανύσει ένα ε, τελείωτο γολγοθά αν θέλετε. Ε, κάπου διάβασα ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μειωθεί το, η περίοδος αυτή στους 12 μήνες. Καταλαβαίνετε δηλαδή στο παρελθόν ο χρόνος αυτός στα κράτη-μέλη ήταν ένα με δύο χρόνια. Τώρα όμως ε, εδώ χρειάζονται μέχρι τρία χρόνια. Βέβαια για κάποια επιχείρηση αυτά τα τρία χρόνια είναι τεράστιο χρονικό διάστημα. Κοστίζουν πολύ και οδηγούν σε πολλές πολυπλοκές. Θα πρέπει η διαδικασία αυτή να ε, ε, απλουστευτεί. Μου φαίνεται ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό γιατί δεν πρόκειται για μια ε, διατάραξη εσωτερικής αγοράς αλλά για καλύτερε δυνατότητες marketing. Όταν έχει κάποιος να προσφέρει ένα ειδικό προϊόν. Και εδώ θεωρώ επίσης ότι θα ήταν καλό να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη ε, το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί τα στάνταρ για τους ελέγχους αυτούς φαίνεται ότι είναι πολύ διαφορετικά και η συχνότητα των ελέγχων επίσης είναι πολύ διαφορετικές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορούσαμε οι έλεγχοι αυτοί να είναι πιο αποτελεσματικές, λογικές, αλλά και βάσει κάποιων συγκεκριμένων προτύπων. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε μία νέα γραφειοκρατία. Νέα έντυπα, νέα έγγραφα, νέα εμπόδια ιδίως για τις ΜΜΕ. Εγώ στράφηκα προς την Κομισιόν γιατί είδα ότι ε, στην Κίνα φαίνεται ότι έχουν πολύ προχωρήσει. Ε, έχουν τώρα παραδείγματο χάρη παραγωγή ε, ζαμπών Πάρμας γιατί ονομάζανε κάποια πόλη ή κομμόπολη στην Κίνα Πάρμα και παράγουν εκεί αυτό το ζαμπόν. Είναι πολύ ευρηματική λοιπόν και θα πρέπει να προσφροντίσουμε να μην έχουμε ε, ζαμπότης πάνω από την Κίνα. Θα πρέπει η Κομισιόν να το λάβει υπόψη στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε αυτές τις χώρες. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Γιατί πια οι καταναλωτές θα μπερδευτούν τελείως. Γι' αυτό υπέβαλα και τη σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν με την παράκληση να ασχοληθούν με το θέμα. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι καλό να συνεχίσουμε με τις ονομασίες ε, γεωγραφικής προέλευσης. Νομίζω κάτι τέτοιο ε, θα πρέπει να είναι βέβαια πιο σαφές και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή και να μειωθούν οι διαδικασίες όπως σας είπα. Πρώτα σε ευχαριστώ κυρία Χολμάγερ. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους θέλει να υποβάλει κάποια ερώτηση. Φαίνεται ότι όχι. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον η Κομισιόν θέλει να αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας πείτε πώς λέγεστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο, την εκπρόσωπο του Ελεκτού αλλά και την κυρία Χολμάγερ που έδειξε πόσο μπορεί να βοηθήσει ο διάλογος, η συνεργασία και η ειλικρίνεια. Ήταν υποδειγματική η συνεργασία και η σχέση μας. Να πω επίσης ότι για μας η άσκηση αυτή ήταν ιδιαίτερα αποδοτική, επικοδομητική και χρήσιμη. Γιατί πήραμε κάποια απόσταση και είδαμε ξεκάθαρα τις ελλείψεις, ε, τις αδυναμίες του συστήματός μας και έτσι μπορούμε πιστεύω να βρούμε και μέτρα και τρόπους να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά. Νομίζω ότι είναι ένας από τους τομείς, ένα από τα θέματα για τα οποία μπορεί κανείς να πει ότι ε, πιο πολλά είναι αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Στόχος κοινό είναι να βελτιώσουμε όλα αυτά τα σημεία, του ελέγχους, τις διαδικασίες και το βαθμό της συνειδητοποίησης, ευαισθητοποίησης παραγωγών και καταναλωτών για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία να πω πρώτον ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη που ήδη κάποιες από τις συστάσεις αυτές είχε συνέχεια. Δηλαδή στα τακτικά σχέδια ελέγχου της Κομισιόν περιλαμβάνονται πλέον οι έλεγχοι για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Να άλλη μια καλή ε, ένδειξη της ε, υποδειγματικής συνεργασίας. Και Έχουμε και το Better Training for Safer Food, καλύτερη κατάρτιση, εκπαίδευση για πιο ασφαλή τρόφιμα. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει ένας καλύτερος έλεγχος όλο αυτό το ε, τομέα. Για το 2012 θα έχουμε πέντε κύκλους κατάρτισης, επειδή βιάζομαστε όμως δεν θα σας πω λεπτομέρειες, απλά σας δω ότι έχει ήδη δρομολογηθεί αυτό το πρόγραμμα. Να πούμε λίγα πράγματα για το μέσο. Ε, τελικά ε, ναι ή όχι. Εμείς είμαστε ε, Τη άποψη ότι δεν χρειάζεται κάτι καινούριο. Απλά πρέπει του κανόνε που έχουμε πρέπει να του εφαρμόσουμε καλύτερα. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Πρέπει λοιπόν να δούμε επιτόπου πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή των κανόνων του κανονισμού 882 και των κανονισμών για τι γεωγραφικέ ενδείξει. Αλλά εν παρόδο να υπογραμμίσω ότι η πρόταση τροποποίηση των κανονισμών 1510 και 1509 που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από την Κομισιόν ε, ουσιαστικά έχει να κάνει με μια διευκρίνηση των υποχρεώσεων των κρατών μελών κατ' ουσίαν. Βέβαια, το λεχθέντος πρέπει να παραμείνουν κάποιες διαφορές γιατί ο αντίκτυπος των γεωγραφικών ενδείξεων, η χρησιμοποίηση του μέσου δεν είναι ίδια ακριβώ ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και τα είδη προϊόντων που είναι, ε, που τυχάνουν αυτής τι ε, προέλευσης επίσης είναι διαφορετικά και έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Πρέπει να πω ότι σημειώνουμε το στόχο και του Κοινοβουλίου και του Ελληνικού Συνεδρίου παρόλα αυτά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τη συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή των ελέγχων. Σε ό,τι αφορά τώρα τι διαδικασίε, πράγματι είναι χρονοβόρε οι διαδικασίε γιατί μιλάμε για προστασία τη πνευματική ιδιοκτησία. Ναι, μπορούμε να το βελτιώσουμε και το έχουμε ήδη ε, ξεκινήσει. Υπάρχει πρόταση για να συντομευθούν οι προθεσμίε όχι μόνο τη Κομισιόν αλλά και των κρατών μελών. Γιατί, θέλω να το πω αυτό αν με επιτρέπετε, πρόκειται ε, για ε, μια κακή παράδοση τη ε, Κομισιόν. Δηλαδή, όταν ε, ουσιαστικά επεκτείνει τι προθεσμίε, το κάνει για να έχει καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και έχει διάλογο για κάθε φάκελο που λαμβάνει για να μην υπάρξει απόρριψη. Θα πρέπει να δούμε και ε, τις διαδικασίες ε, ε, που ισχύουν στα κρατημέλη, που πολλές φορές επιμηκύνονται. Εμείς όταν λαμβάνουμε το παιδί, αν θέλετε, το προϊόν δηλαδή αυτού του ελέγχου, ξεκινάμε και εμείς τον έλεγχό μας, πάρα πολύ αναλυτικό, υπεύθυνο, όπως μας ζητά να είμαστε στις αναλύσεις μας στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναγνώριση εκ μέρους των καταναλωτών και των παραγωγών αυτού του συστήματος. Να πω ότι το σύστημα αυτό πρώτον απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, κατά κύριο λόγο. Η παραγωγή εκεί απευθύνονται στις εθνικές αρχές. Και οι εθνικές αρχές είναι αυτές οι οποίες μας στέλνουν ε, την αίτηση καταγραφής, καταχώρησης. Θα μπορούσε ε, να πει κανείς ότι πράγματι είναι ένα πολύπλοκο σύστημα και υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθεί ο βαθμός αναγνώρισης. Αλλά έχουμε την ένδειξη ότι και εδώ έχουμε βελτιώσει. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε ένα λογότυπο που είναι πλέον υποχρεωτικό εδώ και όχι πολύ καιρό και επίση γιατί η εκθετική αύξηση ε, των αιτήσεων καταχώρησης δείχνει ότι αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα επίση ότι σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχει παράδοση τη γεωγραφική ένδειξη. Τώρα αρχίζει το σύστημα να δει και να γίνεται γνωστό. Κάποιε χώρε ε, κλείνουν πιο πολύ στο εμπορικό σήμα, που είναι μια άλλη, ε, ένα άλλο τρόπο. Παράλληλο με αυτόν τη ε, γεωγραφική ένδειξη. Τέλο, θα ήθελα να αναφερθώ στι ενισχύσει τη κυρία Χολ Μάγερ για το διεθνέ επίπεδο. Μιλήσατε για την Κίνα συγκεκριμένα. Να σα καθησυχάσω. Δεν θα δεχθούμε εύκολα γκολ από την Κίνα, ε, πρέπει να σας πω. Έχουμε ε, βασικές μέρημνες. Πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Πρέπει να προστατευτούν και δικές μας γεωγραφικές ενδείξεις αυτές τις χώρες. Και οι αρχές τρίτων χωρών πρέπει να συμμετάσχουν και αυτές στον έλεγχο των αγορών τους. Και εμείς θα προσέξουμε πάρα πολύ τα πράγματα αυτά. Και αν υπάρχει είτε κάποια απομίμηση, είτε μία παράτυπη ονομασία γεωγραφική ένδειξη, όλα αυτά να τα επισημαίνουμε και να διορθώνονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπενίτε Σάλλας από την Κομισιόν για την τοποθέτησή σας αυτή. Τώρα θα ήθελα να ξαναρωτήσω η κυρία ε, θέλει το λόγο. Να πω κάποια λόγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αποτελεσματικότητα του όλου προγράμματος μπορεί να βελτιωθεί πολύ φθηνά και πιστεύω ότι η έκθεσή μας μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση και για να παίξει τον πρωταρχικό ρόλο για να προστατεύσει τα καταχωρημένα νόματα θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες προδιαγραφές για την πραγματοποίηση των ελέγχων. Αυτό δεν θα πρέπει να αυξήσει πραγματικά τη γραφειοκρατία, αλλά θα βοηθήσει να εξασφαλίσει το ότι το πρόγραμμα θα εξακολουθεί να δικαιολογεί την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές και άλλοι εμπλεκόμενοι και για να εκμεταλλευτούμε περισσότερο το δυναμικό που έχει το σχήμα για την υποστήριξη τη οικονομία τη υπαίθρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει αποτελεσματική στρατηγική, καλύτερη ευαισθητοποίηση και μεγαλύτερη αναγνώριση του λογοτύπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εισηγήτρια, αν θέλει το λόγο, για να ολοκληρώσουμε. Κυρία Χολμάιερ. Νομίζω δεν έχω τίποτα να πω πια. Σας ευχαριστώ απλώς και ελπίζω ότι με τις ονομασίες αυτής προελεύσεως θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο που είχαμε ορίσει στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστώ, ναι. Καλά είναι. Να ακούμε και ότι μια έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου μπορεί να εφαρμοστεί προς σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι καλύψαμε και την καθυστέρηση που είχαμε. Ευχαριστώ και αυτό. Έχει έρθει ήδη ο Αντιπρόεδρος κ. Πιτέλα εδώ. Τον καλωσορίζω με καρδιότητα στην Επιτροπή μας. Και μου λένε ότι ο Γενικός Γραμματέας κ. Βέλες επίσης βρίσκεται καθοδόν. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω μεταξύ μας τον εσωτερικό λεκτό του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, τον Ρόμπερ Κάλβιν. Καλωσορίσατε στο σημείο 12 μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής 2010 πρόκειται να εξετάσουμε τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εδώ μία σειρά ερωτήσεων που υποβάλαμε στον αρμόδιο αντιπρόεδρο και στον γενικό γραμματέα και αυτό σας παρακαλώ στην συζήτηση που θα ακολουθήσει να βασιστούμε σε αυτό το ερωτηματολόγιο. σκοπεύουμε να κάνουμε το εξή. Καταρχήν, θα υπάρχει μια γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου και θα ήθελα να καλωσορίσω από την ευκαιρία μάλιστα και τον κύριο Λούι Καλέα που εκπροσωπεί το ηλεκτρικό συνέδριο. Κατόπιν θα υπάρχει μια σύντομη τοποθέτηση του αντιπρόεδρου κυρίου Πιντέλα και κατόπιν την τοποθέτηση του Γενικού μας Γραμματέα, του κυρίου Κλάους Βέλλερ, προτού δώσουμε το λόγο στον ιστορικό ελεκτή και περάσουμε στη συζήτηση. Με μια δήλωση και ερωτήσεις του εισηγητή μας, του κυρίου Μπογκουσλάβ Λιμπεράτσκι. Έχουμε δηλαδή πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας.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 Λοιπόν κύριε Βέλε, μόλις είπα πώς, τι θα κάνουμε ακριβώς που θα είναι το πρόγραμμα. Θα αρχίσουμε με την τοποθέτηση του ηλεκτρικού συνεδρίου και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκαλέα και να το προσκαλέσω να μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη. Στην έκθεσή μας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ειδική αξιολογήσεως των διοικητικών δαπανών, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στο κεφάλαιο 7, το ελεκτικό συνέδριο κάνει μια γενική αξιολόγηση σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες για όλα τα θεσμικά όργανα και άλλους οργανισμούς ε, ομού. Βεβαίως βασίζουμε την εκτίμησή μας επί των δοκιμών γενικών τυχαίων δειγμάτων συναλλαγών που καλύπτουν όλους τους φορείς. Τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως που διενεργήθη για το 2010 είναι θετικό και το ελεκτικό συνέδριο μπόρεσε να συμπεράνει ότι οι συναλλαγές που οδηγούν στις διοικητικές δαπάνες ε, το 2010 όσον αφορά όλες οι υλικές πτυχές ήταν συναλλαγές νόμιμες και τακτικές με τα χαράς λέγουμε, ότι αυτό ακολουθεί την παρόμοια κατάσταση που επικρατούσε και το περασμένο έτος. Το ελεκτικό συνέδριο κάνει και συμπροματική εργασία για να παρουσιάσει ε, σειρά παρατηρήσεων επί καθενός θεσμικού οργάνου και φορέως. Το συμπληρωματικό έργο που διενεργούμε έχει σαν στόχο επιλεγμένα θέματα. Δηλαδή, υπολογισμό και πληρωμές μισθών, αποζημιώσεων, συντάξεων και διαφόρων ε, δαπανών για τις αποστολές, διαδικασίες ε, προσλήψεων, μονίμου προσωρινού και προσωπικού και προσωπικού επισυμβάση, καθώς και συμβάσεις για προμήθειες. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ελεκτικό συνέδριο κάνει κάποια σχόλια σε σχέση με τους εξής τομείς σχόλια όσον αφορά αδυναμίες όσον αφορά κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται όσον αφορά την υποδοχή ομάδων επισκεπτών καθώς και ότι υπάρχει μεγάλη βάση δίδεται σε πληρωμές σε μετρητά δεν υπάρχει επαρκή δήλωση και διαφάνεια όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού επισυμβάση. Υπάρχουν κάποια κενά όσον αφορά του κανονισμού περί προμηθειών. Υπάρχει διαφορά μεταξύ εσωτερικών κανόνων για την εφαρμογή του προϋπολογισμού που χειρίζονται οι πολιτικές ομάδες και του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα ποσά κατεβλήθησαν στις πολιτικές ομάδες και τέλος ε, περιορισμούς και λήψεων αφορά την αποτελεσματικότητα της εκ των προτέρων επαλήθευσης όσον αφορά κάποιες πτυχές ε, της εκτελέσεως του προϋπολογισμού. Στην έκθεσή μας επίσης ε, σχολιάζουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τις συστάσεις προτέρων εκθέσεων, δηλαδή τη συνέχεια που δίδεται τα σχόλια που, όσον αφορά τη συνέχεια ή follow-up comments. Ένα από αυτά τα σχόλια αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την πληρωμή των κοινωνικών επιδομάτων στα μέλη του προσωπικού, το, Ευρωπαϊκό, το Ελεκτικό Συνέδριο σε πρώτερη έκθεση είχε συστήσει ότι σε κάποια χρονικά διαστήματα θα πρέπει το προσωπικό να παρουσιάσει διάφορα έγγραφα που θα επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση. Το Ελεκτικό Συνέδριο έλαβε υπόψη τα μέτρα τα οποία έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Αυτή είναι η σύνοψη που θεωρούσα ότι αρμόζει στην ευκαιρία αυτή και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαλέα για αυτή την παρουσίαση σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνο για θέματα προπολογισμού, τον οποίο χαιρετίζω μεταξύ μας και του δίνω το λόγο. Κύριε Πιτέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να χαιρετήσω και εσάς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο, όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Χαιρετίζω πολύ εγκάρδια τον κύριο Λιμπεράσκη και του εύχομαι καλή τύχη ε, διότι ανέλαβε το, τη θέση του Κοσμήτωρα. Ξέρετε πολύ καλά, είναι εισηγητή για την απαλλαγή 2010 του Κοινοβουλίου. Και ευχαριστώ και του άλλου και εισηγητή και τον δόκτωρα Λουί Καλέα. Χαιρετίζω επίση που εκπροσωπεί το ελεκτικό συνέδριο που πριν από, πριν από λίγο παρουσίασε τα σχόλια του ελεκτικού συνεδρίου. Όπως υπενθυμίστηκε και σε άλλε ακροασει, όπως υπενθύμησε σε άλλες ακροάσεις, απέναντί σα, Είναι τιμή για μένα που είμαι μέλο τη της Επιτροπής. Είχα την τιμή να ανήκω σε αυτή την Επιτροπή στην πρώτη μου θητεία και έχω έξοχε αναμνήσεις από τη θητεία μου σε αυτή την Επιτροπή. Σήμερα, ως συνήθω συνοδεύω με τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, τον κύριο Βέλε, και τον κύριο Γκάλμπιν, Ρόμπερτ Γκάλμπιν, που συμμετέχουν σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε συγκεκριμένο ερώτημα που ίσως ανακύψει. Όπω γνωρίζετε πολλοί από εσά, είναι τώρα μια συνήθεια η πρόεδρο του Κοινοβουλίου που έχει ευθύνε για τον προπολογισμό να συμμετέχει σε αυτή την ακρόαση. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να τη από την οπτική των καλών σχέσεων και της καρποφόρας συνεργασίας που θέλει να συνεχιστεί ε, το Προεδρείο με την Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού. Στόχο τη ανταλλαγή απόψεων σήμερα είναι να ενημερωθούμε για την εκτέλεση των κονδυλίων που προβλέπονται στον προπολογισμό μα για τι διοικητικέ δαπάνε του 2010 και ε, και τις πιστώσεις που είναι στον προϋπολογισμό και αυτές που απορρέουν αποφάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέτος και που είχαν κάποια συνέπεια όσον αφορά τον προϋπολογισμό θα πρέπει ήδη να έχετε τον κατάλογο των αποφάσεων, άρα αποφεύγω να επαναλάβω αυτέ τι αποφάσει. Θα πρέπει να έχετε λάβει και την απάντηση του Γενικού Γραμματέα στο ερωτηματολόγιο όσον αφορά την απαλλαγή. Πριν δώσω το λόγο στου επόμενου αγορητέ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα στοιχείο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και ε, δίνει σημασία και το Προεδρείο σε αυτό. Δηλαδή διαφάνεια συνεργασία, διάλογος ήταν και παραμένουν σημαντικές σταθερές ε, των εργασιών μας το Προεδρείο από την πλευρά του κάνει προσπάθειες ώστε οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο του προπολογισμού αυτού του θεσμικού οργάνου να ε, φροντίζουν να υπάρχει υγιής διαχείριση και διαφάνεια. Ξέρουμε ότι ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου για προφανή λόγος είναι ο πιο γνωστός προπολογισμό από εμά. Αυτό δεν σημαίνει προφανώς όμως ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει εγγύηση όσον αφορά τη διαφάνεια. Αντιθέτως μάλιστα θα πρέπει να προσέξουμε όμως να μην ε, δείξουμε υπερβολικό ζήλο υπονομεύοντας αποφάσεις που ήδη υιοθετήθηκαν από τις πολιτικές αρχές διότι αυτό θα αντέβαινε το ίδιο το πνεύμα ε, της διαδικασίας της απαλλαγής. Τούτο λεχθέντος θα πρέπει να πω ότι εδώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη στις εργασίες του Γενικού Γραμματέως και των Γενικών Διευθύνσεων που εκπροσωπεί ε, των προσπαθειών που καταβάλουν για τη διαχείριση των εργασιών του Κοινοβουλίου από την πλευρά μας ως αντιπρόεδρος ε, υπεύθυνο για τον προπολογισμό μαζί με τον κύριο Βίταλ είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί, διαθέσιμοι ε, για συνεργασία. Ε, κάθε φορά που θέλετε καλή, οι ερωτήσεις που εμπνέονται από, την, ε, από τον πόθο σας για διαφάνεια και ανοιχτή ε, διαχείριση θα βρίσκουν πάντα μια απάντηση ειλικρινή και ανοιχτή και δίνω τώρα το λόγο στο Γενικό Γραμματέα τον Κλάους Βέλε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για τα τόσα φιλικά λόγια μας είπατε και θα ήθελα πραγματικά να δώσω το λόγο στον Γενικό Γραμματέα να μας κάνει τη δική του έκθεση. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω ευχαριστώντας ε, το Ελεκτικό Συνέδριο για την καλή συνεργασία, όπως και στο παρελθόν, και χαίρομαι που γενικά πήραμε μια θετική έκθεση, παρόλο που βέβαια, όπως πάντα, υπάρχουν τομεί όπου μπορούμε να βελτιωθούμε. Και ευχαριστώ και τον ιστορικό ελεκτή για την καλή συνεργασία. Καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία ε, το οποίο νομίζω ότι βελτιωθήκαμε δομικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 και στο 2011 και μετά να αναφερθώ σε πιο σημαντικά θέματα. Κατόπιν βέβαια θα δοθούν απαντήσεις κατοδελτών και στις μεμονωμένες ερωτήσεις. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι καλή αίτηση ότι το Νοέμβριο του 2011, μέχρι τον Νοέμβριο μάλιστα, δεν υπήρχε τίποτα ανοιχτό, καμία κρίσιμη δράση ανοιχτή από τον εσωτερικό έλεγκτη. Δηλαδή όλες οι συνεργασίες που είχαμε και με τις γενικέ διευθύνσεις ασχολήθηκαν με τις κρίσιμες αυτές δράσεις και αυτό ήταν επιτυχές και έτσι μπορούσαμε να ε, εξαλειφθούν αυτές οι κρίσιμες υποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει πολλά να κάνουμε, όπως το θυμάμαι υπήρχαν 68 υποθέσεις ανοιχτές ε, πάλι μείωση γιατί υπήρχαν 88 το περίσμενο έτος και χαίρομαι που κάναμε μια καλή πρόοδο σε αφορά τη συνεργασία. Δεύτερον, προσπαθήσαμε η εργασία μας μέσα σε πέραση της δημοσιονομικής διαχείρισης να βελτιωθεί μεταξύ άλλων και ε, γενικοποιώντας ε, το θέμα των διευθύνσεων ε, για τους πόρους, δηλαδή εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, έχουμε σε όλες τις γενικές διευθύνσεις μία διεύθυνση για τους πόρους. Έχουν δηλαδή μία δομή, έχουν για τα χρήματα προσωπικό, την πληροφορική και αν υπάρχει ανάγκη στον τομέα της ε, τεχνολογίες πληροφόρησης ε, των κτηρίων ε, και του προσωπικού να μπορούν να συνεργάζονται οι γενικές διευθύνσεις καλύτερα και ελπίζουμε ότι τα πρότυπα στον τομέα αυτό θα μπορέσουν πραγματικά να βελτιωθούν και να αυξηθούν. Και θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω και ένα άλλο διαστρωτικό μέτρο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε όσον αφορά την δημοσιονομική διαχείριση να επανεξετάσουμε γενικά την πληροφορική μας χρησιμοποιώντας ένα software, ένα λογισμικό που ήδη χρησιμοποιεί και το Συμβούλιο και εδώ πρόκειται πάλι για βελτιωμένη διαθεσμική συνεργασία και θέλουμε επίσης να έχουμε και ένα στοιχείο cost accounting, δηλαδή ε, λίγο του κόστους όχι συγκεκριμένο για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ε, τη δυνατότητα προς το, πολιτικό επίπεδο να ενημερώνεται όσον αφορά το κόστος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του κοινοβουλίου και ελπίζουμε ότι αυτό το λογισμικό να υπάρχει στη διαθέσιμο στην αρχή της καινούριας της μελλοντική θητείας. Αυτά κατά γνώμη είναι τρία σημαντικά διορθωτικά μέτρα. Θα μπορούσα ίσως να αναφερθώ και σε τέσσερις μεμονωμένους τομείς. Καταρχήν, η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού το προηγούμενο έτος ήδη μας ε, προειδοποίησαν ότι θα πρέπει να κάνουμε και δομικές εξοικονομήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Δηλαδή, όχι εξοικονομήσεις που θα είναι αποφασιστικές και αποτελεσματικές για ένα χρόνο, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα. Στις διαπραγματεύσεις ε, το περασμένο φθηνόπερο κάναμε τις οικονομίες στον τομέα των, της τη της τάξης των 10 εκατομμυρίων κάθε και της μετάφραση των κειμένων 11 εκατομμυρίων. Αυτό ήταν σημαντικό γιατί ταυτόχρονα βέβαια το Προεδρείο αποφάσισε να αλλάξουμε τον τρόπο εργασία μα. Παραδείγματο χάρη, εάν χρησιμοποιούνται διερμηνεί μετά τα μεσάνυχτα στο Στρασβούργο ε, πρέπει να είναι ελεύθερη την επόμενη ημέρα για λόγους της προστασίας του εργαζομένου. Εάν εργαστούν μετά τις 11 δεν μπορούμε να τους ε, χρησιμοποιήσουμε το πρωί της επομένης. Μια που δεν ξέρουμε όμως ακριβώς πώς θα αρχίσει μια συνεδρίαση, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε διπλή κάλυψη. Και γι' αυτό το η Προεδρία αποφάσισε ότι οι συνεδριάσεις οι συνεδριάσεις της, ε, των Επιτροπών θα τελειώνουμε οπωσδήποτε στις 10 το βράδυ και τις οραμέλες στις 11.30. Επίσης αποφασίστηκε οι επιτροπές να κατανείμουν τις ε, συνεδριάσεις τους καλύτερα ανά την εβδομάδα, δηλαδή να μην συνεδριάζουν οι επιτροπές μόνο Τρίτη και Τετάρτη, αλλά Δευτέρα και Τρίτη ή Τρίτη και Τετάρτη για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους μόνιμους διερμηνείς του σώματος και σας είπα από όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα κάνουμε μια εξοικονόμηση 10 εκατομμυρίων ανά έτος. Και επίσης όσον αφορά τις μεταφράσεις αποφασίσαμε το κρέο να μην το έχουμε ε, σε όλες τις γλώσσες πράγμα που σημαίνει μια εξοικονόμηση 8,6 εκατομμυρίων ανά έτος. Άμα το πολυπλασιάσετε επί μια σειρά ετών θα δείτε πόσα χρήματα είναι αυτό. Θα υπάρχει όμως πάντα σε μια ε, δια, γενικά ε, δευρυμένη γλώσσα. Θα υπάρχει σε, στις νέες τεχνολογίες και αν κάποιος ε, ε, βουλευτής εργαζ... Ε, ιδιαίτερα για κάποιο σημείο, οπωσδήποτε θα το έχει στη διάθεσή του. Αυτές οι εξοικονομήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν άπτονται τις ποιότητες ε, των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους βουλευτές. Και θα ήθελα να σας πω ότι μια καλύτερη συνεργασία με τους γενικούς διευθ... διευθύντες και τους διευθυντές της ε, μετάφρασης και της διερμηνίας έχουμε ένα benchmarking για τους πόρους το 2011 με μεταφορά 100 θέσεων για άλλες, ε, για, σε άλλες υπηρεσίες είναι μια τεράστια εξοικονόμηση που γίνεται κάθε χρόνο έτσι ή μάλλον σε ένα χρόνο έτσι. Και αυτό έγινε και κοινωνικά αποδεκτά με ανοιχτές θέσεις που υπήρχαν και μπορέσαμε έτσι να έχουμε και μια νέα διεύθυνση για τον έλεγχο των επιπτώσεων ή και μια μονάδα για την οικονομική διακυβέρνηση χωρίς να χρειαστεί να ζητήσουμε περισσότερο προσωπικό και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και για την καλή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνίας και Μετάφρασης. Με, αμέσως μετά την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου και μία έκθεση του εσωτερικού Ελεκτή έγιναν επίσης έντονες συζητήσεις στο Προεδρείο για ένα θέμα στο οποίο πετύχαμε σημαντική πρόοδο. Έχουμε μια καλή κατανομή τώρα μεταξύ του κόστου, του, του, του, κόστους για τη μεταφορά για την απόσταση και, το, και του κόστους για την ε, διανυκτέρευση και διατροφή. Έχουμε τώρα για την διανυκτέρευση ένα καταποκοπήν ποσόν 60 ευρώ είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό που δεν μπορεί κανένα να πει ότι στο Στρασβούργο τη Βρυξέλλες μπορεί κανείς να μείνει με λιγότερα λεφτά 40 ευρώ για τη διατροφή και 19 ανά χιλιόμετρο. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά τα ποσά είναι αρκετά χαμηλά και επιτρέπουν επίσης πλήρη διαφάνεια και σαφήνεια στον αφορά το κόστος. Επί σειρά ετών είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολισμού είχα πει ότι εκείνη την ημέρα άνοιξε το παρλαμετάριο γιατί με ρώτησαν πότε είχε ανοίξει αυτό το παρλαμετάριο για τους επισκέπτες υπάρχουν κάποια αριθμητικά στοιχεία βέβαια δεν έχει λειτουργήσει ακόμα ένα ολόκληρο έτο. Ε, θεωρούμε ότι οι επισκέψει θα είναι λιγότερο το χειμώνα από το καλοκαίρι και την άνοιξη. Παρόλο που δεν υπάρχουμε ακόμα, δεν αναφέρεται ακόμα και στους ταξιδιωτικού οδηγούς. Το πρώτο έτος θα έχουμε 250.000 επισκέπτες περίπου στο Παλαμετάριο. Για ένα πρώτο έτος νομίζω το αποτέλεσμα αυτό είναι πάρα πολύ καλό και τα σχόλια που ακούσαμε όσον αφορά και την όλη δομή και προσφορά του Παρλαμεντάριου είναι γενικά θετική. Στα επόμενα έτη, όταν θα γίνει πιο γνωστό και όταν θα εγγραφεί και στο εξωτικούς οδηγούς κλπ, φανταζόμαστε ότι ο αριθμό αυτός θα αυξηθεί. Ένα άλλο θέμα που συζητείται σήμερα είναι το ήχος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Εδώ νομίζω υπάρχει επίσης μια σειρά καλών ειδήσεων Μία πολύ ουσιαστική είναι ότι ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κ. Παρόζο, ανέλαβε την υποχρέωση να συμβάλλει ουσιαστικά από τον κοινοτικό προπολογισμό για τη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει νομίζω ότι αναγνωρίζουν οι, τα άλλα θεσμικά όργανα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κομισιόν, ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που ξεπερνάει τα όρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και γι' αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί και από το Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Αυτά όσον αφορά ορισμένες ε, ε, δομικές ε, διαρθρωτικές αλλαγές και ορισμένα μεγάλα σχέδια. Θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Βέλε, για αυτά που μας είπατε που αντικατοπτρίζουν και αυτά που είχε ζητήσει στο παρελθόν η Επιτροπή μας και ακριβώς στη σήμερα ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την οικονομική απόδοση. Αυτό είναι κάτι που περιμένουν και οι πολίτες που είναι οι φορολογούμενοι. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλβιν, στον εσωτερικό ελεγκτή, να μας δώσει δική του άποψη. Παρακαλώ κύριε Γκάλβιν, έχετε το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, κύριοι βουλευτές, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσω καταρχάς την, πρώτη, την ετήσια μου έκθεση για το 2010. Να πω ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί από τον εσωτερικό ελεγκτή να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο που θα αναφέρει τον αριθμό και το είδος εσωτερικών ελέγχων, τις συστάσει και τις δράσεις που ανελήφθησαν βάσει των συστάσεων. Αντικείμενο τη έκθεσης αυτή απομένων είναι η έκβαση των δραστηριοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών κατά το έτος 2010. Το σημαντικό τμήμα της δραστηριότητας 2010 ήταν η διενέργεια ελέγχων σε διάφορους λειτουργικούς τομείς, ένα ευρύ φάσμα, όπου βλέπουμε την υλοποίηση της διαχείρισης, της δράσης, θα, θα σας δώσω καταρχάς μια σύντομη περιγραφή των αποστολών. Οι εμείς αποζημιώσεις είναι το 20% ε, του συνολικού κόστους μισθοδοσίας και προβλέπεται στο καθεστώς των 2008 2008-2010 ε, κάναμε τον έλεγχο και είχαμε 54 δράσεις για τη βελτίωση των ελέγχων και την εντόπιση συγκεκριμένων κινδύνων. Είχαμε λοιπόν παρακολούθηση των ελέγχων από το 2010, 41 δράσεις, 76% και είδαμε ότι υπήρξε πρόοδος για την μετώπιση ε, σημαντικών τομέων κινδύνου που είχαμε εντοπίσει κατά το παρελθόν. Ωστόσο, βρήκαμε ότι υπάρχει σημαντικό πεδίο ε, για περαιτέρω βελτιώσεις ό,τι αφορά τις διαδικασίες, ε, το περιβάλλον και τις δραστηριότητες ελέγχου, ιδίως ό,τι αφορά την εκχώρηση εξουσιών λήψης αποφάσεων, ενημέρωση και η σύνθεση της μισθοδοσίας με το streamline. Μια άλλη πολύ σημαντική, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι οι δαπάνες σε αποστολές. Είδαμε ότι η ΓΔ προσωπικό και κεντρική διοίκηση υλοποίησαν από τις 22 ε, δράσεις που είχαμε συμφωνήσει. Άρα ε, θα αντιμετωπιστούν από ό,τι φαίνεται τα συστημικά προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει, είχαμε εντοπίσει στην αρχική μας έκθεση. Επίσης υπήρξαν σημαντικές αλλαγές ε, στους εσωτερικούς κανόνες και στα εφαρμοστικά μέτρα που διέπουν τις αποστολές. Και έτσι μετριάσαμε τους δύο βασικούς κινδύνους που είχαμε αναφέρει και μειώθηκε και το κόστος. Ε, μία από τις κριτικές αυτές κρίσιμες δράσεις έχει ολοκληρωθεί και οι άλλοι όχι ακόμη γιατί δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί 100% με τους κανόνες. Αλλά υπάρχει πρόοδος άρα δεν είναι πλέον κρίσιμη. Μεταξύ των άλλων δράσεων πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αποστολών, το ηλεκτρονικό σύστημα και καλύτερη διαχείριση ε, και συμπερίληψη των αποστολών στα στρατηγικά σχέδια. Ζήτησε το 2004 ε, να βελτιωθούν όλες οι συμβατικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Έχουμε έξι δράσεις βελτίωση από το 2008. Η παρακολούθηση από το εσωτερικό ελεκτή δείχνει ότι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μακροχρόνων συμβάσεων και τι κεντρικέ υπηρεσίε, έχουμε καλή εφαρμογή, επιτυχημένη εφαρμογή των δράσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα την τεχνολογία ε, των επικοινωνιών. Σα υπενθυμίζω ότι το 2008 είχαμε κάνει έλεγχο της διακυβέρνησης ε, της τεχνολογίας των ε, επικοινωνιών και είχαμε δει και ποια είναι τα βιομηχανικά πρότυπα. Το αποτέλεσμα ήταν 48 συμπεφωνημένες δράσεις. Στον έλεγχο που κάνουμε το 2010 είδαμε ότι η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ 20 δράσεις της υλοποίησε. Μεταξύ αυτών σημαντικά μέτρα όπως τα συνεργατικά όργανα διακυβέρνησης, έγκριση μιας συνδιάμεσης στρατηγικής για τις τεχνολογίες ICT. Θετικές εξελίξεις που όμως θα είναι αποδοτικές εάν υλοποιηθούν και οι άλλες δράσεις που είχαμε προτείνει. Μεθοδολογία προγραμματισμού, παρακολούθηση των σχεδίων IT, ανάπτυξη δικτών επιδόσεων πλήρης εφαρμογή ενός πλαισίου για την διαχείριση και τον έλεγχο της ασφάλειας, αντιμετώπιση κινδύνων, ιδιοκτησία των ε, διαδικασιών, των δεδομένων, των συστημάτων πληροφοριών. Ο Γενικός Διευθυντής της ε, ITEC με ενημέρωσε πρόσφατα ότι έχει επιτελέσει η υπηρεσία του ε, σημαντική πρόοδο σε σχέση με τις ανοιχτές δράσεις από τότε που δημοσιεύτηκε η έκθεσή μας συμπεριλάβουμε τα νέα στοιχεία στην έκθεση μας το 2012. Μια άλλη σημαντική δράση που ξεκίνησε το 2010 ήταν η του ελέγχου για, τα, για την αποζημίωση της αποδοχής των συνεργατών. Αρχικά στην έκθεση το 2008 είχαν γίνει κάποιε συστάσει. Θέλαμε να δούμε αν εφαρμόστηκαν και ιδίω αν το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι νέε διαδικασίε αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που μα είχαν κάνει να προτείνουμε κάποιε δράσει. Συζητείται η έκθεση των εσωτερικών ελεκτών αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώ θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσει, αλλά μπορώ να σα πω ότι ίσω σε κάποια περιορισμένα θέματα υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω δράση. Πάντω υπάρχει σημαντική εφαρμογή ε, του προγράμματο δράση και να σα πω ότι η υλοποίηση του νέου συστήματο για, την πιστοποιημένη, ε, για του πιστοποιημένου συνεργάτε είναι σε εξέλιξη και θα σας κάνουμε τη σχετική αναφορά το 2012. Περνάω σε άλλους τομείς. Αντικείμενο νέων ελέγχων το 2010. Είχαμε έλεγχο των ομάδων επισκεπτών και της όλης αυτής οργάνωσης. Είδαμε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν, να απλουστευτούν κάποια στοιχεία του ε, συνολικού ρυθμιστικού πλαισίου. είδαμε ότι οι επιδοτήσεις που δίνονται σε ομάδες επισκεπτών υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος μετακίνησης. Αλλαγές επιστηματικονομικές διατάξεις εσωτερικών κανονισμών για την υποδοχή ομάδων επισκεπτών επίσης θα είναι απαραίτητη. Αν θέλει το Κοινοβούλιο να επιτύχει το στόχο του να προσαρμόσει τις επιδοτήσεις με το κόστος το οποίο πραγματικά ε, δαπανάται. Έχουμε διατυπώσει προτάσεις για να έχουμε σαφείς διαφανείς κανόνες για τον υπολογισμό της επιδότησης μετακίνησης, για να μην υπάρχουν ασυνέπειες και διοικητικά προβλήματα. Θέλουμε επίσης να ευθυγραμμιστούν καλύτερα επιδοτήσεις με το πραγματικό κόστος, να υπάρχει καλύτερος καθορισμός των εξόδων που θα επιδοτηθούν, δηλαδή και η διατροφή και η διαμονή. Κατά ε, ποσό. Πρέπει να παραμείνει αυτή η μέθοδος, αλλά να γίνουν και ρεαλιστικές εκτιμήσεις των πραγματικών εξόδων μετακίνησης. Η επιδότηση του, των οδηπορικών σε σχέση και με τον υπολογισμό της καταποκοπήν ε, αυτής ε, δαπάνης, δειγματοληπτική έλεγχη των δικαιολογητικών και παραστατικών είναι ένα άλλο στοιχείο. Και πρέπει να δούμε βέβαια την επιλογή που είχε μελετήσει τότε ο έλεγχος, δηλαδή την πληρωμή σε μετρητά. Να δούμε τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει αλλαγέ στου εσωτερικού κανόνε για τι ομάδε επισκεπτών, κάτι που ενέκρινε στι 30 Νοεμβρίου το Προεδρείο. Και ο έλεγχο του 2012 θα δει πώς αντιμετωπίζουν οι αλλαγές αυτές του κινδύνους που έχουμε εντοπίσει. Το 2010, επίσης, είχαμε τη φάση της υλοποίησης σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού. Και έχει συμπεριληφθεί η έκθεση αυτή στην έκθεση προγραμμάτια του 2011. Θέλαμε να δούμε αν οι αποδοχές δίδονται μόνο σε όσους τις δικαιούνται και αν ε, αντικατοπτρίζεται η αλλαγή στο διοικητικό, στη διοικητική τους κατάσταση με τη μισθοδοσία τους. Εξετάσαμε επίσης την προσέγγιση της ΓΔ προσωπικό για την εφαρμογή σημαντικών μεταβατικών μέσων από τον κανονισμό σε σχέση με τη μισθοδοσία. Είμαστε σε διαβουλεύσεις με τη ΓΔ προσωπικό μετά από το σχέδιο έκθεσης. Έρχομαι στους ε, δημόσιους διαγωνισμούς πέμπτη, πέμπτος ε, έλεγχος ήταν η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ e σε μια σειρά άλλων ελέγχων. Ξεκίνησε το 2010 αυτός ο έλεγχος, αλλά ουσιαστικά το 2011 έγινε η επιτόπου εργασία και τώρα θα αναπτύξουμε τα τελικά μας πορίσματα. Όπως και στους προηγούμενους ελέγχους για τη στρατηγική διαγωνισμών, βασικός στόχος στον έλεγχό μας είναι να δούμε εάν συμμορφώνται γαμα με τις αρχές που διέπουν τις προμήθειες το value for money κυρίω. Και στόχο μα στην περίπτωση τη ITEC ήταν να αξιολογήσουμε την υλοποίηση σημαντικών συμβάσεων πλαισίου που είχαμε εντοπίσει ω ειδικό τομέα κινδύνου κατά το παρελθόν. Άλλα στοιχεία τη δραστηριότητά μα που βλέπουμε και στην ετήσια έκθεση. Έλεγχοι που έγιναν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Είμαστε υπεύθυνοι στο πλαίσιο τη Συμφωνία Διοικητική Συνεργασία για τον Διαμεσολαβητή. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδο. Υπάρχει επίσης περιγραφή του ζητήματος της διασφάλισης της ποιότητας. Πρέπει να τηρούνται τα επαγγελματικά πρότυπα και θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση από εξωτερικού εμπειρογνώμων. Μετά το προπαρασκευαστικό έργο του 9 και του 10 έγινε αξιολόγηση το 2011 και χαίρομαι που σας αναφέρω ότι οι αξιολογητές είπαν ότι είναι ύψιστα τα ποσοστά συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν έλαβα καμία οδηγία, καμία καθοδήγηση που να ε, υπονομεύει την ανεξαρτησία μου και την αυτονομία μου. Θέλω να ευχαριστήσω το Προεδρείο, τον Γενικό Γραμματέα και να ευχαριστήσω για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που ε, παρήχαν όλοι οι διατάκτες στον εσωτερικό ελεγκτή. Σα ε, ε, Σας ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, στον συνάδελφο Λιμπεράτσκι. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αξιότιμη αντιπρόεδρε Πιτέλα, κύριε Βέλε, κύριε Γκαλέα, Κύριε Βαρβίν, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνεται να συζητήσουμε την αποτελεσματικότητα της εκτελέσεως του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010. Και κύριε Βέλε, σας ευχαριστώ εσάς και τις υπηρεσίες σας για τις πληροφορίες ε, που δώσατε στην Επιτροπή μας. Ήταν αρκετά ικανοποιητικές. Αναγνωρίζω ότι πολλά από τα θέματα που θίγονται στις γραπτές ερωτήσεις ξεπερνούν το έτος 2010. Θέματα τα οποία αφορούσαν ειδικά το Κοινοβούλιο. Όμως, είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε πληροφορίες για ευρύτερα ζητήματα και άλλα χρονικά πλαίσια ευρύτερα. Ευχαριστώ το Γενικό Διευθυντή, τους Γενικούς Διευθυντές και το προσωπικό που μας δώσανε και πληροφορίες στις συνεδριάσεις. Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε το ευρύ πεδίο εργασιών που γίνονται στο Κοινοβούλιο. Οι εργασίες αυτές εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινοβουλίου και αναφερόμαστε στο δικό μας θεσμικό όργανο. Καθήκον μας εδώ είναι να εξετάσουμε το θέμα της απαλλαγής του προπολογισμού του 2010 εστιάστηκα ε, στο συγκεκριμένο έτος για την εκθεσή μου. Όμως γνωρίζω ότι οι παρόντες συνάδελφοι θα ήθελαν να θέσουν ευρύ φάσμα ερωτήσεων στη σημερινή συζήτηση και προσβλέπω στο, στη διεξαγωγή ανταλλαγής απόψεων. Σημειώνω το βασικό θέμα που εθίγει σήμερα, τα βασικά θέματα Στο ερώτημά μου θα καλύψω τρεις στοιχές. Πρώτα πολλά, ποσοστά εκτελέσεις του προπολογισμού εν γέννη και στις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Δεύτερον, τομείς υπό εσωτερικό έλεγχο και παρακολούθηση. Τρίτον, πιο συγκεκριμένα θέματα που θα ήθελα να τα απαριθμίσω. Πρώτα, εκτέλεση προπολογισμού. 96% των τελικών ποσών για το έτος εκτελέστηκαν που δεσμεύτηκαν και η χαρτογράφηση μη χρησιμοποιηθέντων ποσών για τα ποσά υπολογίστηκε στο τέλος του 2010. Η προσέγγιση βοηθά τη διαφάνεια και την απαλλαγή. Δεν Πρέπει να αποκρινθούμε από τη χαρτογράφηση, από τις σημαντικές μεταφορές ποσών, ε, να μετακινηθούμε από εκεί και να πάμε στην πλέον διαφανή διαχείριση των ποσών που πάνε στα κτίρια. Δεύτερον, το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Είναι σημαντικό το έργο για να λειτουργεί καλύτερα ο φορέας. Όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Μετά τον έλεγχο που έγινε το 2010 προτάθηκαν κάποια πράγματα. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις διαδικασίες διακυβερνήσεως δικήσεως των γενικών διευθύνσεων. Τι σημαίνει αυτό και ποιες εξελίξεις έλαβαν χώρα το 2011 αναφέρονται. Το θέμα των δαπανών, των αποστολών εξετάστηκε. Πολλές δράσεις χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά την τεκμηρίωση των αποστολών. Χρειάζονται σχέδια για συγκεκριμένες δραστηριότητε. Να δούμε τι πρόοδος μπορεί να ή επετεύχθη και τι απομένει. Τρίτον, συγκεκριμένο, το πρώτο συγκεκριμένο. Κόστος για την ασφάλεια. Έχουμε διαφορετικά στοιχεία για το 2010 από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε γραπτές ερωτήσεις και σε σχέσεις με, με τα στοιχεία που μας δόθηκαν τις συζητήσεις. Υπήρξαν κάποια γεγονότα που έλαβαν χώρα πέρσι και πρόπερσι όσον αφορά την ασφάλεια Χρειαζόμαστε λεπτομέρειες για τις δαπάνες στην ασφάλεια. Θα διευκόλυνε την απαλλαγή. Θα ήταν καλό να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ετησίω από τούδο και στο εξή. Έτσι θα μπορούσαμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της νέας έννοιας της γενικής ασφάλειας. Τι συμπληρωματικές πληροφορίες θα μπορούσαν να προσταθούν για τις προμήθειες. και εκεί που γίνονται διαπραγματεύσεις χωρίς να πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ε, για, την, ε, για τις προμήθειες. Κάπου είχαμε αυξήσει του κόστου σε κάποιε γενικέ διευθύνσει, κάπου μειώσει. Γιατί υπάρχουν διαφορέ, ποιο ο λόγο, τι μπορεί να γίνει. και να χρησιμοποιούνται λιγότερο οι έκτακτες διαδικασίες προμηθειών στις γενικές διευθύνσεις. Το δημογραφικό βάρος δεν αναφέρθηκε πουθενά μέχρι τώρα. Οι διάφορες επικότητες στο προσωπικό του Κοινοβουλίου. Σαν Πολωνός, χαίρομαι που τα νέα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται καλά στο προσωπικό. Κυρίως στο μέσο και χαμηλότερο επίπεδο. Υπάρχει όμως σαφής υποεκπροσώπηση από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν περισσότεροι Βέλγοι και Λουξεμβούργοι από ό,τι θα αναμενόταν αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος των ελόγων χωρών. Πώς μπορεί να διορθωθεί η ανισορροπία και πώς μπορεί να πετύχει την αλλαγή το Κοινοβούλιο. Παραμένει αυτό το ερώτημα. Äh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιγητά, κύριε Λιμπεράτσκι, για την αποθέτησή σας και για την ερώτησή σας. Θα έλεγα τώρα, καταρχήν έχουμε ένα γύρο των πολιτικών ομάδων και μετά ένα δεύτερο γύρο με άλλους συναδέλφους. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Α, στην κυρία Ιβάνοβα για το ΕΛΚ. Δύο λεπτά να περιοριστεί ο καθένας αν είναι δυνατόν. Θα κάνω ό,τι μπορώ, λέει κύριε Ιβάνοβα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν τα σύντομα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο κύριο Πιτέλα και τον Γενικό Γραμματέα, το ε, Ελεκτρικό Συνέδριο και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, καθώς επίσης και τον εισηγητή για τη συνεργασία του. Καταρχήν έχω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που πήραμε πλήρες απαντήσει απαντήσεις στις γραπτές μας ρωτήσεις έγκαιρα φέτος. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Βλέποντας τις απαντήσεις βλέπουμε ότι στα πιο σημαντικά τμήματα έχει επιτευχθεί η πρόοδο. Τα πιο σημαντικά τα ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας, η πρόεδρο στην πληροφορική, τις προτάσεις για εξοικονομήσεις στο τομέα της μετάφρασης και της διερμηνίας κλπ. κλπ. Βέβαια πάντα μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. λόγω του περιορισμένου του χρόνου, θα αναφερθώ σε λίγους τομείς που θεωρώ ότι είναι κρίσιμοι και πάρα πολύ σημαντικοί. Καταρχήν ασφάλεια. Υπήρχε μια δήλωση ότι κατόπιν της ε, ε, διάρρηξης του ταχυδρομείου πέρσι έγιναν πολλά αλλά μέχρι στιγμής εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πραγματική διαφορά στον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας. Μπορείτε να μας δώσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αλλαγής που επετεύχθη για να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια στο κοινοβούλιο. και στην βελτιώσει και ποια θα είναι τα απτά αποτελέσματα αυτού της ιδέας. Δεύτερον, οι δημόσιε προμήθειε αναφέρθηκε και από το ηλεκτρικό συνέδριο και από τον εισηγητή. Αυτά είναι θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και τη διαχείριση τη διαδικασία. Θέλω να σα ρωτήσω ποια θα είναι τα μέτρα που θα αναβληθούν για το θέμα αυτό και κατά πόσο ορισμένε μονάδες που ξεχωριστά εργάζονται στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Πώς θα φροντίσετε να πετύχετε όμως συνεργασία ε, διαφάνεια και λιγότερο ρυθμό σφαλμάτων που φαίνεται ότι είναι προβληματικό ε, μετά όσον αφορά το θέμα των ομάδων επισκεπτών και αυτό ήταν κάτι που έθιξε και το ηλεκτρικό Συνέδριο και ο Συντορικός αλλά θα ήθελα να στραφώ τώρα στον Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θεωρείτε ότι τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από το Προεδρείο τον Νοέμβριο του περασμένου έτους θα βοηθήσει πιο διαφανές σύστημα και θα μειώσει το κίνδυνο υπερβολικών πληρωμών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ, ιδίως που ήσασταν τόσο σύντομοι. Ο Γιάννη Μιούλτερ, από την άλλη, αν θέλει. Eh, eh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αλλάξω. Μια μιλάω αγγλικά, μια θα μιλάω ολλανδικά ο εισηγητής ε, και ο κ. Ε, παρακάλεσε να αναλάβω τις δικές του ερωτήσεις που θα τις υποβάλω στα Ολλανδικά. Πρώτο ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοβουλία της Άλτε σε μια σειρά ψηφισμάτων και σε αυτό για το προβλησμό 2012 ζήτησε αξιολόγηση του προπολογισμού. Παρ' όλο αυτό δεν έχει γίνει τίποτα. Πώς πότε πρόκειται να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Δεύτερον, γιατί δεν εφάρμοσε πάντα το Προεδρείο συστάσεις του Κοινοβουλίου που εμείς είχαμε ζητήσει σε σώμα. Παραδείγματο χάρη το βραβείο για τους δημοσιογράφους. Άμα δείτε τις απαντήσεις του Γενικού Γραμματέα, βλέπετε ότι το Προεδρείο δεν εφαρμόσει το την ψήφισμα αυτό του σώματος. Και μια τρίτη ερώτηση. Κοιτάω γύρω μου και δεν βλέπω σχεδόν κανέναν που δεν έχει κάποιο ηλεκτρονική συσκευή μπροστά του. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσαμε όλα τα έγγραφα να τα μεταβάζουμε μόνο ηλεκτρονικά. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα γινόντουσαν τεράστιες εξοικονομήσεις χαρτιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Äh, äh, ευχαριστώ κύριε Μούλτερ, ο κύριος Στάς. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, και εγώ θα μιλήσω Ολλανδικά. Πάντα μιλάω Ολλανδικά στο κάτω-κάτω. Εκτός αυτού, στην καμπίνα περιθμών 5 υπάρχουν ε, κάποια άτομα που έχουν την ευκαιρία τώρα να ξεκουραστούν λίγο. Γιατί όταν μιλάω Ολλανδικά δεν χρειάζεται οι διερμηνείς της Ολλανδικής καμπίνας να εργαστούν. Καλό είναι και αυτό που και που. Υπάρχει ένα σχέδιο που αφορά τις ηλεκτρονικές επιτροπές της, ή e όπως λέγονται και εκεί όλα τα έγγραφα μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά. Μπορεί κανένας να τα κοιτάξει στον υπολογιστή του, να προωθήσει και τις τροπολογίες κλπ. Γίνεται αυτό δηλαδή ήδη, αλλά το ερώτημά μου είναι διαφορετικό. Κύριε Βέλε, αναφερθήκατε στο Παρλαμεντάριο. Καταπληκτική πρωτοβουλία με μεγάλη επιτυχία από ό,τι μου λένε. Αλλά πήραμε και πολλά έγγραφα όσον αφορά το κόστος ε, του ε, οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Γιατί δεν συνδέθηκαν αυτές οι δύο πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι χάσαμε εκεί τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Γιατί υπήρχε μεγάλο κόστος για το παραμετάριο και το ίδιο κόστος θα το υπομισθούμε τώρα για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Χάσαμε μια ευκαιρία νομίζω. Τώρα. Είμαι πολλά χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο. Σημάμαι τον κύριο Ντάνκερτ που ήταν ο δεύτερος ε, πρόεδρος του Κοινοβουλίου το 1983, 84 Είχε ένα ιστορικό γραφείο με πέντε συνεργάτες. Πέντε. Σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή και ο Γενικός Γραμματέας έχει ένα πολύ μεγαλύτερο εσωτερικό γραφείο. Ξέρω βέβαια ότι ε, έχει και περισσότερα πράγματα να κάνει, αλλά παρόλα αυτά είναι ε, κρυκτική αυτή η αύξηση. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κάτι να βελτιωθεί. Γιατί καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι άτομα που ήταν στο εσωτερικό γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Προέδρου, κάποια στιγμή χρειάζεται να έχουν κάποια άλλη θέση στο οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου. Μήπως έτσι υπάρχει κάποια, ε, κάποιο κίνητρο να ε, ε δοθούν ε, ε, κάποιες προαγωγές Μήπως γι' αυτό υπάρχουν τελευταία τόσες πολλές ε, διευθύνσεις και χρειαζόμαστε άρα τόσους πολλούς διευθυντές. Μήπως είναι αυτή η τάση ότι άτομα που ήταν στο, στο εσωτερικά γραφεία των, του Πρόεδρου κλπ. που είναι πολύ ικανοί άνθρωποι, δεν λέω, δεν το αρνούμε, τώρα αναλαμβάνουν κάποια διεύθυνση ως διευθυντές. Ε, πρόεδρος. Η κυρία Ανδρεάσιν έχει το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις του Προεδρείου του Γενικού Γραμματέα, του Εσωτερικού Ελεγκτού, των Ελεγκτών. Θα αναφερθώ σε κάποιες πτυχές των ερωτήσεων. Ερωτήσεων όπου είναι ασαφείς οι απαντήσεις, για να πω το λιγότερο. Ερώτηση 1, παραδείγματι. Λένετε ότι έγιναν δίπλωση 182 θέσεων ανακατάταξη δεν μας δίνεται εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται αυτό το εγχείρημα. Σε απάντηση του ερωτήματος 2 λέτε ότι πρόκειται να αντικαταστήσετε το λογισμικό για τα διοικητικά έγγραφα, το GDA. Το κόστος δεν λέτε τίποτα. Ερώτηση 3. Ρωτούμε αν οι δράσεις που προτείνει ο εσωτερικός ελεγκτής εφαρμόστηκαν. Ουδεμή απάντησης. Δεν γνωρίζουμε. Ανέφερε ο εσωτερικός ελεγκτής ότι στην περίπτωση του τομέα πληροφορικής μόνο 20-40 προταθήσεις δράσεις εφαρμόστηκαν. Κατά τα λοιπά δεν γνωρίζουμε. Ερώτηση 4. Δεν υπάρχει ένδειξης ποια τεχνική υποστήριξης παραμένει λειτουργούσα μεταξύ των συνόδων στο Στρασβούργο. Ερώτηση 27. Ρωτήσαμε ποιο είναι το κόστος των αποστολών. Και δεν έχουμε απάντηση. Πότε θα μπορούσαμε να έχουμε απάντηση. Το επίμαχο θέμα για μένα. Πρέπει να το αναφέρω προσεκτικά γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι δίνω νούμερα στους δημοσιογράφους Ευρωπαϊκό Οίκο ιστορία, ο Οίκο ευρωπαϊκή ιστορία. Κύριε Βέλε, μας δώσετε καλά μαντάτα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μοιραστεί το κόστο. Λυπούμε που λέγω, και το είπα και προηγουμένω, αυτά δεν είναι καλά μαντάτα. Ο ίδιο φορολογούμενος πληρώνει το κόστο του οίκου Ευρωπαϊκή Ιστορίας. Το ότι μοιράζεται το κόστο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημαίνει τίποτα, ο φορολογούμενος την πληρώνει. Άρα δεν είναι καλέ ειδήσει για μένα. Θα ήθελα να έχω σαφή ορισμό, καθορισμό των δαπανών, του κόστους. Σελίδα 12 γίνεται σύγκριση μεταξύ του αρχικού σχεδίου, του επιχειρησιακού και ακολούθων. Και αναφέρεστε σταθερό και μεταβλητό κόστος. Θα ήθελα διαχωρισμό αναφέρεστε στο βασικό προσωπικό, πανεπιστημιακό, αυτά τι θεωρούνται μεταβαλλόμενο κόστος, σταθερό, πάγιο κόστος. Πώς γίνεται η κατανομή μεταξύ πάγιου και μεταβλητού κόστους και άλλων δαπανών. Θα πω αυτό που είπε και ο Μπαρτ Στάς. Δεν συμφωνώ ότι το Παρλαμεντάριουμ και ο, Ευρωπαϊκός, ε, ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα έπρεπε να συνδυαστούν. Εγώ πιστεύω δεν θα έπρεπε να υφίστανται, να υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κύριε Αντρέασεν, ο κύριος να έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα για τις απαντήσεις που έδωσε. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε μέσω οικονομικής κρίσης και κάθε μέρα έχω αλληλογραφία από πολίτες που ανησυχούν για το κόστος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά τις απολαβές των βουλευτών. Εκτός από την επιστροφή του το κόστος μετάβασης, υπάρχει ε, εκτός λέω από το κόστος διαμονής και ε, ημερησίων δαπανών υπάρχει και ένα κόστος που πληρώνεται για την μεταφορά. Ίσως να μπορείτε να μου πείτε κάτι παραπάνω σε αυτά. Ίσως αυτές οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται μόνο βάσει αποδεκτικών στοιχείων γιατί αλλιώς παραμένει αυτή η εικόνα ότι εμείς ε, ξοδεύουμε ό,τι θέλουμε. Κατάλληλα, οι προτάσει που γίνουν για τον επόμενο προβλησμό είναι καλές, ε, κάποια αξιολόγηση νομίζω είναι σωστές. Και τώρα για τον οίκο της ε, Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ήδη ο κ. Μούλντε το ανέφερα. θα πρέπει να δει κανένας αυτή τη μελέτη της νομικής υπηρεσίας που είναι δύσκολο να την πάρει κανένα στα χέρια του. Μια μελέτη που λέγεται ότι εάν το θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα χρήσης μιας ε, νομικής φάσης, αλλά δεν λέει τίποτα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του οίκου αυτού. Θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν για την εφαρμογή κάποιων μέτρων και δεν ξέρω κατά πόσον είναι δυνατόν να αποφευχθούν στις προλήψεις, να προληφθούν, προσληφθούν ε, μέλη οικογενειών. Εγώ βλέπω ότι όταν έχει, ε, έχουμε αυτή την, ε, τη δική μας εκπομπή στη τηλεόραση, κάποιες λίγες χιλιάδες ακροατών μονάχα παρακολουθούν. Πώς δεν θα μπορούσαμε να τα μεταδώσουμε μέσω κοινών καναλίων για να μην έχουμε ε, το συμπληρωματικό έξοδο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάτι να αλλάξει εδώ. Πρώτα σε ευχαριστώ κύριε Τιγιού. Ολοκληρώσαμε τώρα το γύρο των πολιτικών ομάδων και θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις πριν περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ή μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους δύο βουλευτές. Ε. Ο κύριος Έτελε έχει αριστεί το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους κύριους Πιτέλα και Βέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση με παρουσία σας εδώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι Υπήρξε πρόοδος εδώ στο Κοινοβούλιο, σημαντική, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. There is no mopping up. Only two uh, transfers. Του mopping up, της ε, σάρωσης. Τα ποσά των μεταφορών είναι τεράστια. Το ίδιο είναι τελικά transfer και mopping up κατά την άποψή μου. Μάλλον κακή πειθαρχία ήταν ε, να σταματήσει αυτή η διαδικασία και το ίδιο περίπου είναι και οι μεταφορές, αυτές, αυτά τα εμβάσματα. Οπότε δεν ήταν αυτή η ιδέα που είχαμε εμείς προτείνει να αντικατασταθεί το ένα σύστημα από το άλλο. Να έρθω τώρα στο θέμα της ασφάλειας. Εγώ τουλάχιστον ορατές αλλαγές δεν έχω δει. Η ασφάλεια βέβαια δεν είναι πάντοτε ορατή. Έχει πιαστεί κανένας από την αστυνομία για ε, τη ληστεία αυτή. Βρήκαν κάποιον. Και κάτι να κάνετε με τη θέρμανση, γιατί έχουμε ξεπαγιάσει εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ. Ναι, τώρα το κατάλαβα ότι κάποιοι κρυώνουν και γι' αυτό είχαμε έτσι την ημερησία διάταξη για να μπορέσει ο γενικό γραμματέα να είναι παρόν ναι, και να αρχίσει να κρυώνει και ο ίδιο. Και ε, εκτό ε, πρακτικών, θα ήθελα να σα πω ότι ω νέο ε, πρόεδρο έχω προετοιμάσει ε, μια πορτοκαλάδα έξω. Εάν προτιμάτε βέβαια ε, σαμπάνια θα μπορούσατε να το κάνετε αν θέλετε σύμφωνα με την παράδοση. Πραγματικά κάνει κρύο εδώ μέσα, έχετε δίκιο, αλλά ίσως μπορέσουμε να αντέξουμε μέχρι το τέλος και να το λύσουμε στο μέλλον. Ίγκες σκρέσλα έχει το λόγο. Κοιτάξτε, τίποτα πιο βαρύ θα ήθελα, νομίζω, για να μπορέσει να με ζεστάνει. Η πορτοκαλάδα τι να κάνει. Τώρα, όσον αφορά αυτό το θέμα των ομάδων των επισκεπτών, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Θα ήθελα να ακούσω κάτι παραπάνω και θα ήθελα μάλιστα αυτό, αυτός ο έλεγχος να υπάρχει στην αίθουσα ασφαλών εγγράφων, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον καθένα. Σήμερα τις προφορίες που έχω ε, άκουσα ότι με την ε, σε ρευστό πληρωμή για τις ομάδες των ε, επισκεφτών το Κοινοβούλιο είναι αντίθετο με τις οδηγίες για το πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Πρώτος, ωραία, θα ακούσουμε τώρα Γενικό Γραμματέα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μία-μία σε ερωτήσεις. Αλλά όταν υπήρχαν περισσότερες της μία ερωτήσεις για κάποιο θέμα, θα μου επιτρέψετε να τις απαντήσω από κοινού. Καταρχήν, όσον αφορά τις ερωτήσεις του εισηγητή και του δημοσιονομικού προγραμματισμού. Τα τελευταία χρόνια μπορέσαμε να έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα εκτέλεσης, από ό,τι κατάλαβα και υψηλότερα από ό,τι τα άλλα θεσμικά όργανα. 96% και καμιά φορά μάλιστα και 97% μέχρι και 98%. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται να έχουμε 100 ε, και 101% γιατί δεν επιτρέπεται να εργαστούμε με πιστώσεις. Πρέπει πάντα να μείνουμε κάτω από τη ε, γενική, από τη γενική πρόβλεψη γιατί δεν επιτρέπεται να πάρουμε δάνειο. Και γι' αυτό το 96, 97, 98% νομίζω ότι είναι πολύ καλά στοιχεία. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη σας ερώτηση για την πολιτική σχετικά με τα κτίρια. Μπορεί κανείς να δει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος με την μεσοπρόθεσμη πολιτική για τα κτίρια. Αυτό ήταν ένα σημείο που είχε θυγεί πολλές φορές, πολλά χρόνια από την Επιτροπή Προπολογισμού και υποθέτω και ελέγχω του προπολογισμού, ότι θα πρέπει να υπήρχε κάποια διαφάνεια όσον αφορά τις προθέσεις και τις ανάγκες στον τομέα της πολιτικής για τα κτίρια και ότι το Προεδρείο θα έπρεπε να διευκρινίσει την κατάσταση. Τώρα έχουμε το ίμιση θητείας πίσω μας, ε, μπορούμε να κάνουμε δηλαδή κάποιο απολογισμό και έχω να πω ότι πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν για τη μεσοπρόθεσμη πολιτική για τα κτίρια πραγματικά έτσι γίνονται. Δηλαδή η αγορά ορισμένων κτίριων που χρησιμοποιεί το ε, το κοινοβούλιο προς το κτίριο Μοντουαγέ και το κτίριο Ρεμάρα. Τα συμπληρωματικά 30.000 τετραγωνικά που χρειαζόμαστε στις ε, Βρυξέλλες. Έχουμε το λεγόμενο επίσης κτίριο B που το αγοράζουμε τώρα όπως αποφάσισε το Συμβούλιο να το αποκαλέσει σύμφωνα με το όνομα του Βακταφ Χάβελ ένα κτίριο που χρησιμοποιήθηκε και από το Συμβούλιο και από εμά και ήταν πολύ καλή αυτή η συμβουλική απόφαση που ελήφθη. Λοιπόν, η στρατηγική για τα κτίρια που αρχικά ακούγεται σαν μια αφηρημένη έννοια, βήμα προς βήμα, κομμάτι προς κομμάτι ε, πραγματοποιείται. Δηλαδή εκεί έχουμε ένα καλό πλαίσιο δράσης όχι μόνο για το Προεδρείο αλλά και για τις Επιτροπές Προπολογισμών και Έλεγχου του Προπολογισμού. Και εδώ θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Συνέδριο πολλά χρόνια στο παρελθόν μας είπε ότι εάν κάποιος μακροπρόθεσμα θέλει να χρησιμοποιήσει ένα κτίριο δεν είναι πολύ οικονομικός τρόπος να νοικιάζει. Είναι λοιπόν σπατάλη των πόρων και μας είχε πει το Ελεκτρικό Συνέδριο να μην νοικιάζουμε, να αγοράζουμε τα κτίρια και ακολουθούσαμε το Ελεκτρικό Συνέδριο αν θυμάμαι καλά, το 8% μόνο των και αναγκών μας ε, νοικιάζουμε και το 92% μας ανήκει. Εξοικονομούμε λοιπόν 163 εκατομμύρια νίκη το χρόνο γιατί έχουμε αγοράσει κάποια κτίρια. που πρέπει βέβαια να χρησιμοποιούμε μια που τα έχουμε. Και η διαδικασία που ειδωτήσαμε τώρα με μεμονωμένες μεταφορές που επιτρέπει στην Επιτροπή Προπολογισμού να κάνει μια αξιολόγηση, να πει ναι, να πει όχι, είναι μια πιο διαφανής διαδικασία αυτή και να μην έχουμε μια σφαιρική μεταφορά μόνο πόρων. Όσον αφορά την δομή διακυβέρνηση στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, το 2010 είχαμε εφαρμόσει μια μεγάλη μεταρρύθμιση γιατί χωρίσαμε τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού σε τρεις διευθύνσεις και οι ουσιαστικές μεταφορές ε, πόρων ε, συγκεντρώνονται στην διεύθυνση Β. Αυτό μας δίνει μια καλύτερη δυνατότητα να εργαστούμε επαγγελματικά και να αποφύγουμε ελλείψεις και σφάλματα. Εκτός αυτού, αυτό που ήταν και αντικείμενο του ελέγχου του ιστορικού λεκτή, ήταν σε ποιο επίπεδο λαμβάνονται ποιες αποφάσεις στην διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά πόσον υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι στις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Γιατί βέβαια είναι σαφές ότι εάν ληφθεί μια απόφαση η οποία επαναλαμβάνεται πολλές φορές ακόμα και μικρά ποσά λόγω της επανάληψης έχουν σημαντικές επιπτώσεις και γι' αυτό είναι καλό που έχουμε μία επαρκή ε, αρχή ελέγχου και η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων στην διοίκηση και ενδεχομένως και στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν χρειάζεται. Από την άλλη μεριά όμως αυτό σημαίνει ότι δεν έχει νόημα το ανώτερο επίπεδο να επιβαρύνεται με συνεχείς αποφάσεις ρουτίνας. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να βρούμε τη σωστή απάντηση σε αυτό που μας σύστησε και ο ιστορικός συλλεκτής. Όσον αφορά τις ε, αποστολές του προσωπικού, καταρχήν είναι αξιολογό ότι οι αποστολές μεταξύ των τριών τόπων εργασίας μειώθηκαν σε ένα χρονικό διάστημα δύο ετών. Αν θυμάμαι καλά, από 14.100 σε 11.400. Είναι σημαντική μείωση αυτή των ε, επαγγελματικών αυτών ε, ταξιδιών που δεν είναι τυχαία, είναι θελούσια. Εξετάστε δηλαδή ποιος θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταβεί κάπου Βέβαια αυτό είναι και μια επίπτωση της κατάστασης γραφείων και χώρου στο Στρασβούρο που δεν επιτρέπεται να παίρνει κανένα πολλού συνεργάτε μαζί του. Έχουμε λοιπόν εδώ μια θετική εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όταν, συμβιβάζεται, όταν συμπληρώνεται συγγνώμη, ε, η εκαθάριση του ταξιδίου, πρέπει τώρα να αναφέρει κανένας αν είχε και κάποιον ε, συνταξιδιώτη στο αυτοκίνητό του και κατά πόσον ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κατοικείται από ένα άτομα ή από περισσότερους του ενός. Δεν θέλουμε να είμαστε αδιάκριτοι, αλλά και αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις ε, δημοσιονομικές. Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε τακτικά κατά πόσον είναι δυνατόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία τηλεδιάσκεψη αντί μία μετάβαση. Μετά. Ε, αναφέρονται δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι το πραγματικό στοιχείο των υποχρεώσεων και το άλλο είναι αυτό που είχαμε προβλέψει. Ευτυχώς οι πραγματικές υποχρεώσεις είναι χαμηλότερες από τη βάση ε, στον προπολογισμό. Ε, οι δεσμεύσεις αυτές ήταν 47,5 προγραμματισμένες και 43,9 πραγματοποιήθηκαν. Γι' αυτό έχετε αυτή τη διαφορά αυτών των στοιχείων στο έγγραφο. Το ένα είναι η βάση στον προπολογισμό και το δεύτερο είναι η πραγματική, τα πραγματικές δαπάνες. Επίσης αναφέρθηκε θετικά ότι ο αριθμός των των χορηγήσεων μειώθηκε από 89 το 2009 το 2010 σε 49 μόνο σχεδόν δηλαδή το ίμιση αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα έτη είχαμε την ανησυχία ότι θα έχουμε μια συνεχή αύξηση. Άρα δεν για αυτό το 2010 μειώθηκε κατά το ίμιση. Ρωτάτε γιατί. Για δύο λόγους κατά βάση. Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 χρειάστηκαν αυτές τις διαδικασίες παραδείγματος χάρη για να μπορέσουμε γρήγορα να αντιδράσουμε στις απαραίτητες εργασίες με την πτώση της οροφής ε, της αίθουσας της Ολομερίας στο Στρασβούργο. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει κάθε χρονιά και γι' αυτό ήταν αυτό το 2000 ένα έκτακτο κόστος και επίσης ήταν και οι δαπάνες για την προετοιμασία των ευρωεκλογών και γι' αυτό τώρα μειώθηκαν οι δαπάνες αυτές. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι υπάρχουν και πολύ λογικές ε, αιτίες για αυτές τις διαδικασίες. Παραδείγματος όταν έχουμε στην αγορά μονοπολικές καταστάσεις. Αν υπάρχει ένας μόνο που προσφέρει την υπηρεσία αυτή, ίσως είναι καλό να έχουμε και αυτή την διαπραγματευτική διαδικασία. Η έκτη ερώτηση αφορούσε το κατά πόσον έχουμε αρκετούς συνεργάτες από κάποια κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε στην ε, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Μεγάλη Βρετανία και γιατί έχουμε δυσκολίες σε αυτές τις χώρες. Βέβαια δεν έχουμε ποσοστώσεις στο Κοινοβούλιο, αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τώρα κάποιες διαθροτικές δυσκολίες. Το πρώτο είναι ότι με το νέο καθεστώς που σε ισχύ το 2004 η αρχική πληρωμή μειώθηκε πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή έχουμε 3-4 ε, βαθμούς ε, που είναι χαμηλότερη από την παλιά αρχική εισαγωγή. Και βέβαια όταν εγώ τον διαχωρισμό, ο, ο διαγωνισμός αυτός προκυρήσεται στο πιο χαμηλό επίπεδο. Βέβαια σε ορισμένε χώρε δεν υπάρχει πρόβλημα να ε, ε, ε, προβλέψουμε τη δυνατότητα προσλήψεων από τις χώρες αυτές από άλλε χώρε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, από τη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματο καταρχήν γιατί η κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια λέει ότι δεν χρειάζεται στα σχολεία να μαθαίνουν γλώσσε τα παιδιά. Αλλά οι υπάλληλοι χρειάζεται να ξέρουν δύο ξένε γλώσσε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λίγοι Βρετανοί που έχουν δύο γλώσσε στην κατοχή του. Εκείνοι που ξέρουν δύο γλώσσε προέρχονται από διπλωματικέ ε, οικογένειε ή έχουν ζήσει στο εξωτερικό όποιος έχει όλα τα, όλα τα προσόντα. Δηλαδή έχει δύο ξένες γλώσσες, ξέρει δύο ξένες γλώσσες, έχει ένα καλό ε, δίπλωμα και λοιπά, δεν πάει στις Βρυξέλλες βέβαια, θα εργαστεί στην City του Λονδίνου και ε, κερδίζει πολύ περισσότερο. Δεν είμαστε λοιπόν ανταγωνιστικοί εκεί. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν πολύ καλή νομοθεσία, παραδείγματος χάρη για τις γυναίκες όσον αφορά την προστασία μητρότητα. Στην Σουηδία, παραδείγματο χάρη, εγώ είδα πολλέ φορέ ότι υποψήφοι, γυναίκε υποψήφοι από τη Σουηδία απόστεναν την υποψηφιότητά τη ή δεν δέχτηκαν την προσφορά όταν έμαθαν όλους τους όρους πρόσληψης, όχι μόνο το μισθό δηλαδή, αλλά παραδείγματο χάρη και την κοινωνική προσφορά στον τομέα της μητρότητας κλπ. Λοιπόν, έχουμε κάποια κράτη-μέλη όπου με τις εισαγωγικούς ε, μισθούς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Σε άλλες χώρες, ναι. Dann Ivanova Κατόπιν, η κυρία Ιβάνοβα αναφέρθηκε στα μέτρα όσον αφορά την ασφάλεια. Καταρχήν θα σας πω ότι και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα που τίθεται από πολλούς και απαντάται διαφορετικά από διάφορους βουλευτές. Ποια είναι η μορφή της ε, ε, ασφάλειας που θέλουμε να έχουμε στο Κοινοβούλιο. Πάνω σε αυτό υπάρχουν πολύ διαφορετικές απαντήσεις. Ορισμένοι λένε όλα θα πρέπει να είναι ανοιχτά και ελεύθερα και δεν θέλουμε καθόλου ελέγχους. Άλλοι λένε ότι η έλεγχη θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να επιτευχθεί συνένεση. Ποια μορφή ασφάλεια θέλουμε να έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προερχόμαστε από μια κατάσταση στην οποία η έννοια ασφάλεια στο Κοινοβούλιο δεν είχε τόσο ύψιστη σημασία. Τώρα στο Πρόεδρο συμφωνήσαμε πάνω σε μια σειρά μέτρων να κλείσουμε λοιπόν τα αδύναμα σημεία Στο παρελθόν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτά. Ε, είχαμε το θέμα του γκαράζ, του, του, του, γκαράζ του Προέδρου και η ενιαία εφαρμογή προτύπων ασφαλείας επίσης. Ένα πρόβλημα ήταν ότι η ασφάλεια στην ε, είσοδο του τύπου ήταν πολύ πιο χαλαρή από ότι στην κύρια είσοδο και γι' αυτό χρησιμοποιείται και αυτή η είσοδος του τύπου. Επίσης, ο έλεγχος των θέσεων των ε, φωτογραφικών και τηλεοπτικών μηχανών που θα δίνουν τώρα καλύτερες εικόνες στο μέλλον, αποφασίσαμε να μειώσουμε κάπως την, ε, τους εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή ο έλεγχος και η επιτήρηση στον τομέα της ασφάλειας δεν θα γίνεται από εξωτερικούς συνεργάτες πια. Δηλαδή η επιτήρηση των ε, ε, αρμοδίων για την ασφάλεια δεν μπορεί να δοθεί σε εκείνους που μας διαθέτουν το προσωπικό αυτό. Όχι, αυτό θα πρέπει να γίνεται από δικό μας προσωπικό. Και όσον αφορά την ε, ε τον έλεγχο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν το κοινοβούλιο, θα πρέπει να γνωρίζουν τους βουλευτές κλπ. Γιατί η εξωτερικοποίηση, αν θέλετε, που δεν γινεται ποιότητα, στο τέλος τέλος δεν είναι φτηνότερη, είναι πιο ακριβή. Το Προεδρείο επίσης αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές ζώνες ασφαλείας στο κοινοβούλιο. Δηλαδή δεν μπορούν όλα να είναι εξίσου ασφαλή, αλλά παραδείγματος χάρη στον τομέα του ε, μη κυκλίου, των γραφείων του Προέδρου ή των βουλευτών χρειαζόνται υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας από ότι στο κάτω, στο διάδρομο που υπάρχουν τα διάφορα ε, καταστήματα ή που υπάρχει και καφετέρια. Αυτές είναι κάποιες ιδέες και προσανατολισμοί που υιοθέτησε το Προεδρία και που θα εφαρμόζονται σιγά σιγά και που ήδη εν μέρη εφαρμόζονται. όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Στην τελευταία μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού αποφασίσαμε να μην υπάρχει πια κεντρική ευθύνη αλλά κάθε γενική διεύθυνση να είναι αρμόδια για το δικό της τομέα. Αυτό βέβαια σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα έχουν και την ευθύνη την οποία δεν επιτρέπεται να τους πάρουμε. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να δώσουμε εμείς κεντρικά είναι οι συμβουλές και αυτό το κάνουμε μέσω του λεγόμενου Procurement Forum του Βήματος για τις ε, Προμήθειες. Εκεί δίνουμε τις συμβουλές, αλλά ο καθένας που είναι υπεύθυνο για τις εντολές δεν μπορεί να απαλληφθεί της ευθύνης του. Και γι' αυτό εκεί που υπάρχουν έντονες υψηλές δαπάνες έχουμε δημιουργήσει συγκεκριμένες μονάδες που επιτρέπουν αυτή την άσκηση της αρμοδιότητας. Αναφερθήκατε επίσης στις ομάδες των επισκεπτών. Είχαμε έντονες συζητήσεις στο Προεδρείο. Μία σειρά μέτρων ήδη υιοθετήθηκαν ιδίως ο διαχωρισμός των διαφορών ε, χρημάτων που δίνονται και νομίζω ότι τα χρήματα αυτά είναι τώρα ε, έτσι ούτως ώστε να είναι ρεαλιστικά γιατί νομίζω το 60, τα 60 ευρώ για διανυχτέρευση στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο δεν είναι υπερβολικό ποσό 40 ε, για την διατροφή επίσης δεν είναι υπερβολικό ποσό ούτε τα 19 ανά χιλιόμετρο νομίζω όσον αφορά τις πληρωμές είδος αποφασίσε διαφορετικά το ε, Προεδρείο από εκείνο που είχε προταθεί και λόγους, για λόγους πρακτικούς και μετά από έντονες συζητήσεις. Ο κύριος Μούλτε αναφέρθηκε στο θέμα των μελετών ε, αξιολόγησης και εξοικονόμησης ε, πόρων. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι καμιά φορά κανείς αναθέτει μια μελέτη, καλύτερα θα να κάνει την εξοικονόμηση από πριν. Αποφασίσαμε λοιπόν να μην κάνουμε καμία μελέτη που θα παρουσιάζεται μετά από ένα έτος, αλλά να κάνουμε αμέσως την εξοικονόμηση 21 εκατομμύρια όσον αφορά τις γλώσσες Φιλιππίν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο. Και επίσης μεταφορά των θέσεων των ε, υπαλλήλων, σας είπα 100 ε, κατά τη διάρκεια του 2011 που πήρανε μετάθεση εσωτερική Νομίζω ότι έτσι αποδείξαμε ότι μπορούμε να βρούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα και μπορούμε να κάνουμε τις εξοικονομίες αυτές γλίγορα, με συνέπεια και χωρίς να χρειαζόμαστε μελέτες. Η σχέση τώρα του Προεδρείου και με την Ολομέλεια. Βέβαια το Προεδρείο εξακολουθεί να παραμένει υπεύθυνο για την αξιολόγηση. Η ομάδα εργασίας επικοινωνίας εξετάζει προσεκτικά το θέμα των βραβείων Στι τελευταίε συνεδρίε του Προεδρείου είχαμε έντονη συζήτηση γι' αυτό και το γεγονό ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση. Αλλά η διαδικασία τη εξέταση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά έγγραφα, ο Μπαρτστά με βοήθησε δικαίω ε, γιατί πραγματικά έχουμε το πρόγραμμα που λέγεται ηλεκτρονικό κοινοβούλιο ή Parliament και είναι σαν ένα πρόγραμμα πιλότο σε κάποιες επιτροπές. Ο στόχος είναι μέχρι θητείας να υπάρχουν σε όλες οι επιτροπές τουλάχιστον οι τεχνικές προδιαγραφές να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς χαρτί. Τώρα, κατά πόσον ο κάθε βουλευτής θέλει να εργαστεί χωρίς χαρτιά, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμάς η ευθύνη μας ως, ε, διοίκηση είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, εάν το θέλουν οι βουλευτές. Ο Μπάρτ Στάς αναφέρθηκε επίσης ε, στο νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Κατά πόσον δεν θα έπρεπε να έχει συνδεθεί και συνδυαστεί με το κέντρο των επισκεφτών. Η κυρία Ανδρέα αν έχει ακριβώ την αντίθετη άποψη. Το Προεδρείο είπε θέλουμε για το 2014 να έχουμε μια κοινή εμπειρία από το κέντρο επισκεφτών που έχει σαν επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας που δεν είναι βέβαια εστιασμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά στην ιστορία της Ένωσης της Ευρώπης και να υπάρχει ε, μία, ε, μία δυνατότητα επίσκεψης στο ε, Παλαμετάριο, στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και στην Ολομέλεια συνδυασμένα. Δηλαδή προσπαθούμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες μία εμπειρία που θα συνδέει τα τρία αυτά πράγματα μεταξύ τους. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου μας είπε επίσης ότι υπάρχει νομική βάση εάν το ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ενσωματωθεί πραγματικά στη, στο πρόγραμμά μας για τους επισκέπτες. Τα συμβουλευτικά όργανα είναι πραγματικά συμβουλευτικά και η αρμοδιότητα της απόφασης είναι στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι και αυτό νομίζω σημαντικό. Όσον αφορά τα εσωτερικά γραφεία του, του Προεδρέου και του Γενικού Γραμματέα, βέβαια έχουν κάποια, κάποια μέγεθο, αλλά βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγαλώσει εδώ μεταξύ από την εποχή του κ. Τάνκερ. Έχουμε 6.000 υπαλλήλου μαζί με του υπαλλήλου των πολιτικών ομάδων και συνολικά 11.000 συνεργάτε έχουμε ένα προπολογισμό της τάξης 1,7-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και η δυνατότητα κεντρικών ε, ελέγχου. Ας πούμε και οι τακτικές απαντήσεις ε, προς την επιρροή ελέγχου του προπολογισμού χρειάζεται κάπου να ε, βρουν μια κεντρική ένα κεντρικό σημείο στο από το οποίο θα προέρχονται. Εμείς ε, πέρσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε χωρίς να υπάρχουν συμπληρωματικές ε, προσλήψεις και χωρίς ε, ας πούμε στο παρελθόν όλοι οι τμήματάρχες παίρναν το βαθμό α3 δηλαδή σήμερα θα ήταν α14 τώρα αυτοί οι άνθρωποι σε μεγάλο ποσοστό περνάνε στη σύνταξη και μπορέσουμε να καλύψουμε τις θέσεις αυτές χωρίς προαγωγές και εκεί δηλαδή έχουμε εξοικονομήσεις, είμαστε πιο ορθολογικά οργανωμένοι, χωρίς να δημιουργούμε συμπληρωματικό κόστος. Προς την κυρία Σεν, η οποία έθεσε μία σειρά ερωτήσεων, έχω να πω τα εξή. Καταρχήν όσον αφορά την ε, μετάθεση αυτή των ε, συνεργατών. Αυτή η μετάθεση των 182 συνεργατών δεν κόστησε τίποτα γιατί πρόκειται για θέσεις που υπήρχαν ήδη στο οργανόγραμμα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ανοιχνεύουμε πού δεν χρειάζονται κάποιες θέσεις ε, πια και τις χρησιμοποιούμε αντί να ζητάμε νέες προσλήψεις. Λοιπόν, έχουμε αναφέρει 182 θέσεις για 5 χρόνια και το 2011 ακόμα περισσότερο βρήκαμε θέσεις οι οποίες δεν χρειάζονται εκεί που βρίσκονται αλλά χρειάζονται ίσως κάπου αλλού ίδιος για την ε, πολιτική ενημέρωση των βουλευτών που θα πρέπει να είναι το κεντρικό μας έργο χωρίς να δημιουργηθεί συμπληρωματικό κόστος. Επίσης αναφερθήκατε στο ΚΕΝΤΑ, δηλαδή στο σύστημα διαχείρισης ταχυδρομείου και ε, αρχείων, ετέθη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προβλησμού το ερώτημα κατά πόσον η επεξεργασία μα του θέματο αυτού είναι ιδανική. Εγώ απαντώντας είπα ότι δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή, αλλά ότι χρειαζόμαστε ένα βελτιωμένο σύστημα λογισμικού για να δούμε κάθε φορά πού βρίσκεται κάποια διαδικασία, ποιε είναι οι προθεσμίε κλπ. Δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά ακόμα, δεν μπορώ να σα δώσω στοιχεία, αλλά αυτό το έλλειμμα που αναφέρατε το αναγνωρίζω και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης η κυρία Ανδρέασεν αναφέρθηκε στους εσωτερικούς ελέγχους. και στις ανοιχτές δράσεις. Εγώ είχα πει εισαγωγικά ότι ε, στην ημέρα προθεσμίας δεν είχαμε καμία κρίσιμη ανοιχτή δράση. Είναι πολύ καλή η είδηση αυτή. Και οι άλλες ανοιχτές ε, δράσεις μειώθηκαν από τα 88 στις 68. Καλή η τάση είναι αυτή και δείχνει επίση ότι η συνεργασία με τι γενικέ διευθύνσει για φέτος τουλάχιστον ήταν καλή. Όσον αφορά τις ε, αποστολές αναφέρθηκα, όσον αφορά τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας νομίζω ότι βλέπετε ξεκάθαρα την κατανομή του κόστου σε τρεις τομείς ε, από τα έγγραφα που έχετε. Καταρχήν το κόστος κατασκευής αναφέρονται περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, το κόστος για τον εξοπλισμό. Δεν θέλει κανένας να έχει ένα γιαπί δηλαδή, αλλά πρέπει να έχει σωστή μορφή. Εδώ έχουμε 21 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Τα, αρχικά, τα ακριβή στοιχεία τα έχετε στα έγγραφά σας και μετά τα, οι τρέχουσες δαπάνες, όπου σε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Υπολογισμών και μετά στο Προεδρείο, αποφασίσαμε να μειώσουμε, να ανοίγουμε έξι μέρες και όχι εφτά, να μειώσουμε το προσωπικό, να χαμηλώσουμε τους βαθμούς πρόσληψης του προσωπικού αυτού και να ανανεώνουμε όχι κάθε 8 χρόνια αλλά κάθε 10 χρόνια. Έτσι μειώσαμε το κόστος των, της τρέχουσας δαπάνης δηλαδή και έχουμε τη δέσμευση του κυρίου Μπαρόζο επίσης ότι η Κομισιόν θα θέλει να συμβάλλει. Αυτό βέβαια είναι σωστό, δεν πρόκειται αυτό για διευκόλυνση του Ευρωπαίου φορολογούμενου, αλλά πρόκειται για την αναγνώριση ότι το, ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι σημαντικό μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά για όλα τα θεσμικά όργανα, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον. Ο κ. Δεγιόν αναφέρθηκε στο καταποκοπήν ποσό για την απόσταση ταξιδιών. Αυτό είναι κάτι που ε, διακανονίζεται στο ίδιο το, καθεσ... τον ιστορικό κανονισμό. Αυτό είναι θέμα δηλαδή που θα πρέπει να υποβληθεί στο νομοθέτη και όχι <clears throat> στο εφαρμοστικά όργανα, δηλαδή είναι τμήμα των αποφάσεων που υιοθετούνται μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και μόνο ο νομοθέτης, οι νομοθέτες μάλλον μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους και να το αλλάξουν ούτε το Προεδρείο ούτε η διοίκηση του Κοινοβουλίου. Για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας αναφερθήκατε στη μελέτη. Η μελέτη αυτή ε, κατέδειξε κάθαρα ότι έχουμε μια νομική βάση, αλλά την νομική βάση αυτή την έχουμε μόνο εφόσον ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ενταχθεί μέσα στην πολιτική μας για τους επισκέπτες. Έχουμε 100.000 ε, επισκέπτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε έτος και ζητήσαμε σε κάθαρα τα συμβουλευτικά όργανα να είναι συμβουλευτικά όργανα και η αρμοδιότητα από λήψη απόφαση να είναι στα χέρια του Προεδρείου και αυτό προσαρμόστηκε βάσει της ε, έκθεσης της ε, νομικής Τώρα, όσον αφορά την απασχόληση μελών οικογενείας. Το Προεδρείο αποφάσισε στην περασμένη θητεία θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 5 ετών, η οποία λύγει στα τέλη της ε, θητείας του 2014. Μετά δεν θα υπάρχει δηλαδή καμία βάση για την απασχόληση μελών της οικογένειας. Όσον αφορά το, την τηλεόραση WebTV υπάρχει το θέμα ότι οι εικόνες που παρουσιάζονται εκεί και τα στοιχεία υιοθετούνται πολλές φορές, αναλαμβάνονται από μεγάλες ε, εταιρείε ε, τηλεόρασης για την λεγόμενη δήλωση του Προέδρου State of the Union 200 από ό,τι μου είπανε άλλες ε, υπηρεσίες και κανάλια την αναμετάδωσαν. Έχουμε δηλαδή πολύ σημαντικές έτσι, ε, ε, συνολικά φαινόμενα. Το κόστος μειώνεται από 9 στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Ιταλά αναφερθήκε στις ε, γενικές μεταφορές. Ε, είπα κάτι, το να το ζητήσαμε μεμονωμένες ε, μεταφορές για να μπορεί ε, το Επιτροπή Ελέγχου του Προεπλογισμού να κρίνει κατά πόσο θέλει να την εγκρίνει την κάθε μεταφορά ή όχι. Για την ασφάλεια επίσης αναφέρθηκα όσον αφορά τώρα την θερμοκρασία εδώ στην αίθουσα τι να σας πω. Και εκεί ίσως υπάρχουν διαφορετικές επιθυμίες. Ίσως αν ήταν πιο ζεστή η θερμοκρασία δεν θα ήταν πολύ οικολογική Ο κύριο Στάς παραδείγματος δεν θέλει να ανεβάσουμε θερμοκρασία τη αίθουσα. και ολοκληρώντα, έχω να πω ότι λυπούμε ότι δεν υποβληθεί ερώτηση για το, ε, τη συσκευή αυτή που κόβει τα λαχανικά ε, ε, στο Στρασβούργο. Εγώ ήθελα να σας δείξω ότι αυτό είναι ένα έγγραφο που ένα, μια, ένα μηχάνημα που χρησιμοποιεί φρέσκα λαχανικά για 3.800 γεύματα. Λαχανικά που προέρχονται από τη γύρω περιοχή, άρα δεν ε, και πολύ ε, διοξείδιο δεν παράγεται, συγγνώμη, πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Πρώτα σας ευχαριστώ για την τόσο αναλυτική σας αυτή παρουσίαση. Ίσως ε, οι υπηρεσίες εδώ θε, θεώρησαν ότι είναι μια ψυχρή επιτροπή, η Επιτροπή ελεύθερου και αυτό δεν χρειάζεται πολύ ζέστη. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα θέλω να δώσω στον εισηγητή τον κύριο Λεμπεράτσκι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο ε, γιατί έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν. Δεν ξέρω αν πρέπει να καταβάλουμε χρήματα για υπερορίε στους διερμηνεί. Θέλω να ευχαριστήσω τους κυρίους ε, Καλέα, Κάλβιν και Βέλε για τι επιπρόσθετες πληροφορίε που μας έδωσαν σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου μου, τα μέλη της Επιτροπής, ε, για τα ερωτήματα που έθεσαν για τη συμβολή τους στην όλη συζήτηση. Να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους κοιόδης συζητητές. Κυρίες και κύριοι, η συνεργασία σας μαζί μου είναι μια πραγματική ευχαρίστηση για μένα. Αλλά, χωρίς να θέλω να είμαι αγενής, υπάρχει ε, κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Κύριε Βέλε, είπατε ότι η υλοποίηση του προπολογισμού δεν μπορεί να υπερβεί το 100%. Όμως, λάβαμε μια πληροφορία από τον κύριο Ντε πλήρωσε 30.000 ευρώ συμβολή για το Ευρωκοινοβούλιο. Αν όλοι μας το 2012 πληρώσουμε 30.000 ευρώ, μπορεί να πάρετε το 120 100% συν 100 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Μήπω αυτό θα ήταν μια λύση. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λιμπεράσκη. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο κύριο Πιτέλα και τον Γενικό Γραμματέα Κλάου Βέιλε, καθώ επίση τον εσωτερικό ε, ελεκτή του κύριο Γκάλφιν και όλη την ομάδα του κυρίου Καλέα από το ελεκτικό συνέδριο. Έχουμε ολοκληρώσει εδώ τις εργασίες συνεδρίασή μα. Μία ανακοίνωση έχω να κάνω. 26 Ιανουαρίου του 2012 είναι η επόμενη μας συνεδρίαση. Θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Συνεδρίαση των συντονιστών. Και 9 Φεβρουαρίου του 2012 είναι η επόμενη συνεδρίαση. Πέρα συνεδρίαση.